Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start. Συναδελφοί, ας ξεκινήσουμε. Αύριο έχουμε και το μάτς. Απόψε, απόψε. Έχουμε το Βέλγιο-Γαλλία που φαίνεται ότι είναι σημαντικότερο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ο Πρωθυπουργό του Βελγίου θα πάει στη Ρωσία να δει το παιχνίδι αντί για την ε, σύνοδο του ΝΑΤΟ και να δει τον κύριο Τραμπ. Μια διπλωματική λύση υποθέτω. Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές. Ε, Πρόφορουν το Brexit. Η πρόταση δηλαδή για τις ε, ποσοστώσεις ε, μεταξύ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από το Brexit και τον λόγο έχει η κυρία Κουίστχαουτ Ρόβολ που... για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι Έχουμε πολύ συναρπαστικά θέματα με το Brexit ε, για την ε, τηλεόραση σε σχέση με το Γαλλία, Βέλγιο και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι όμως η πρώτη φορά που ασχολούμαστε συγκεκριμένα με τα τεχνικά ζητήματα γιατί το Brexit ε, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι λανθασμένη απόφαση αλλά θα γίνει και θα υπάρχουν συνέπειες σε όλους τους ε, τομείς εμείς ε, το λέμε αλλά έχουμε την εντύπωση ότι και στις δύο πλευρές της μάχης το ξέρουν, αλλά δεν ε, φαίνεται να τους απασχολεί το ότι θα έχει κάποιες ε, συνέπειες και ότι πλησιάζει. Τώρα λοιπόν, όπως είπα, για πρώτη φορά η Κομισιόν ε, προτείνει έναν κανονισμό για την ε, κατανομή των ποσοστώσεων στον ΠΟΕ μετά από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και για την ε, αλλαγή του κανονισμού 32 2000 του Συμβουλίου. Πολύ τεχνικό το ζήτημα, μπορεί να σας τα πει η Κομισιόν καλύτερα από εμένα πως δηλαδή θέλει να κατανείμει αναλογικά τις ε, ποσοστώσεις. Μου έδωσαν το παράδειγμα των βερίκοκων. Λοιπόν, το θέμα το εξής, εάν τώρα τα βερίκοκα σε σχέση, ας πούμε, αν είχαμε τους 28 θα, παραμείνα, θα παραμέναμε στα ίδια. Εάν λοιπόν από μια ποσόστοση 100 εκμεταλλευτούμε μόνο τα 60 και από τα 60 ε, είχαμε μια σχέση 12-48 θα γίνει μια αναγωγή για να καταλήξουμε στα 100 είτε εξαντληθεί η ποσόστοση είτε όχι. Εντάξει, λογικό φαίνεται αυτό και τώρα να σας πω το εξής. τι θέλω να σου πω. Το... Γιατί και το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα υπάρχουν στα εκτιμώντας. Όλα τα άλλα είναι λογιστικά. Είναι πάρα πολλά νούμερα που αφορούν πάρα πολλά πράγματα στα οποία να σας λέω νομοθετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μπορούμε να δεχτούμε τους αριθμούς αν συμφωνήσουμε με τις αρχές. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε θα ήταν, αν ε, έχει κάποιος την όρεξη, να καθίσει και να προτείνει ένα εναλλακτικό σχήμα. Και έτσι θα μπορούσαμε με βάση την νομοθετική μας εξουσία να προτείνουμε έναν διαφορετικό αλγόριθμο και να πάμε μετά στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και να αποφασίσουμε ότι αυτή η μέθοδος υπολογισμού που προτείνουμε εμείς είναι καλύτερη. Εγώ κάποτε είχα σπουδάσει φυσική και μου φαίνεται κάπως λογικό αυτό το οποίο λένε. Αν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό το οποίο μοιάζει κάπως με νομοθεσία θα έπρεπε να μπει στο ε, διατακτικό στα άρθρα και να γράψουμε έναν αλγόριθμο Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ θυμήθηκα το διδακτορικό μου με αυτούς τους μαθηματικούς ε, τύπους. Να μας δείξει λοιπόν η Κομισιόν τους αλγόριθμους όπως κάνει και το Facebook για να είμαστε έτσι στην ε, επικαιρότητα. Έτσι κάπως ηρωνικά τα λέω αυτά, αλλά ε, νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν. Θα συζητήσουμε πάλι ή φορά σε ποιο βαθμό θα έχουμε πράξεις κατεξιοδότηση και εφαρμοστικές ε, πράξεις ε, και θεωρώ ότι για μια πρώτη συζήτηση ε, αυτά επαρκούν ως βάση. κάτι άλλο έχω να πω ελπίζω πραγματικά να μην έρθει με αυτήν την α, ε, μορφή και να βρούμε μια πιο ανοιχτή έτσι, και λογική λύση αλλά γνωστόν αυτό δεν είναι δικό μας ε, θέμα. Σας ευχαριστώ. David Martin από τους Σοσιαλδημοκράτες. Thanks, Bernd. As you say, on behalf of Alessia and perhaps in some σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μιλώ ε, βέβαια και στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Κάποιος εχθές του ότι ε, ζητάμε συγγνώμη από την Ιταλία γιατί ξεκινήσαμε το καλοκαίρι κλέβοντας τον καιρό σας, ε, το, μετά συνεχίσαμε κλέβοντας το ποδόσφαιρό σας και τώρα τελευταία κλέβουμε και το είδος της πολιτικής σας. Ε, ίσως η Κομισιόν λοιπόν όντως πρέπει να αρχίσει τις προετοιμασίες και λογικά η θέση ε, θα πρέπει να είναι αυτή το κατήγορο. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, πρώτη ερώτηση είναι προς τους Ευρωπαίους εταίρους και την απάντησή τους σε αυτό. Αρκετοί έχουν εκφράσει ε, σοβαρές ανησυχίες. Η Νέα Ζηλανδία πρότεινε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη ενιαία αγορά ως ενιαία αγορά. Γιατί αν και η νέα ρύθμιση θα βασιστεί στην ιστορική χρήση, η μελλοντική χρήση βεβαίως δεν σημαίνει πως ε, ε, είναι εγγυημένη. Οπότε θέλω να συνεχίσουν να διατηρούν την ευελιξία και δεν ξέρω αν έχετε ελέγξει αυτό το είδος την προσέγγιση. Επίσης, ε, κάποιος άλλος μου πρότεινε σε σχέση με το πώς λειτουργεί ο ΠΟΕ, ότι θα ήταν σωστό να έχουμε μια σωστή νομική μορφή, αλλά στην πράξη κάτι τέτοιο δεν θα κάνει διαφορά στην, στην πράξη. Τίποτα δεν θα αλλάξει ε, στον ΠΟΕ, αν δεν κάνουμε τίποτα. Και θέλω να ξέρω αν η Κομισιόν ε, συμμερίζεται αυτή την άποψη. Αυτά και ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η Έμα Μοκλάρκιν από το ECR. Καλημέρα, συνάδελφοι. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα χρειαζόταν και πάλι να περιγράψουμε ε, την θέση της Βρετανικής κυβέρνησης, αλλά Brexit θα πει Brexit και συμβαίνει, θα γίνει δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα όλων αυτών των προγραμμάτων. Η ομαλή ε, εξέλιξη για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βρετανία είναι ο μόνος τρόπος να καθησυχάσουμε τους εταίρους στο ΠΟΕ ότι θα συνεχιστούν τα πράγματα ως έχουν σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει τώρα στον ΠΟΕ και θα έχουμε δηλαδή μια ομαλή μετάβαση. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ένωση θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα ώστε να αποσυνδεθεί από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσπαθήσει να προκαλέσει τη μίνιμουμ ε, διαταραχή και θα να συνεχίσει τις σχέσεις και το εμπόριο με τις τρίτες χώρες ε, φυσικά. Ε, το ECR καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν ε, γιατί η μεθοδολογία που ακολουθεί είναι η πιο δίκαιη για τη Βρετανία και την Ένωση αλλά και για τους εμπορικούς μας εταίρους και ε, χρησιμοποιούνται οι πρόσφατοι οι πρόσφατες ροές στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπολογιστούν αυτές οι υποχρεώσεις. Τώρα, πώς υπολογίζεται ο ακριβής υπολογισμός του ποσοστού χρήσης μιας συγκεκριμένης ε, TRQ ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση. Και το κομμάτι της μη πληρούμενης ε, TRQ μέσω αυτού του μαθηματικού τύπου μπορεί να υπολογιστεί και αν και αυτό, ε, το, αυτό το είδος υπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι κάνει ό,τι μπορεί σύμφωνα με το άρθρο GATT 28 ε, σε αυτές τις προματεύσεις Προσβλέπουμε λοιπόν ε, τις προτάσεις του εισηγητή ώστε να έχουμε μια ομαλή, όπως είπα, μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν βλέπω άλλη εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με την πρόταση. Παρά τη διατήρηση των ποσοστώσεων που έχουν ε, οι διάφορες χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την άλλη αυτό το οποίο ε, καταναλώνεται στην κάθε χώρα. Οι αριθμοί αυτοί υπάρχουν, δεν χρειάζονται περίπλοκες ε, φόρμουλες ή αλγόριθμοι. Για την ΚΟΕ, Χέλμοντ Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ θα έλεγα ότι, όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί να δεσμευτούμε προς τις, σε σχέση με τις υπάρχουσες ποσοστώσεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι κανείς έντιμος με τους άλλους εταίρους με τους οποίους υπάρχουν ήδη συμφωνίες ή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είναι αυτά τα ποσά ρεαλιστικά, είναι σε θέση Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένες αλυσίδε προϊόντων, ε, να διατηρήσει τις ποστώσεις αυτές με τους ε, εταίρους της από τις τρεις ε, τις χώρες. Για παράδειγμα, η συμφωνία με την Ανατολική, με την Τανζανία εκεί όπου υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες ε, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάποιες επιμέρους ε, περιπτώσεις και να εξετάσουμε το θέμα αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάικλ ε, διευθυντής ε, της ε, Διεύθυνσης της Καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε όλοι, η πρόταση είναι κομμάτι του πακέτου, η οποία αποτελείται από δύο προτάσεις. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει την αρμοδιότητα της Επιτροπής να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και μας έδωσε την έγκριση το Συμβούλιο, άρα θα ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ πολύ σύντομα. Αλλά Επίσης, ε, κάναμε μια δική μας ανάλυση και εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και δεν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να πάρουμε το δικό μας ε, ε, δρόμο και να διαπραγματευτούμε μονομερός τις ποσοστώσεις αυτές με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά τα οποία άκουσα σήμερα, δηλαδή το ότι είπατε ότι η μέθοδος την οποία επεξεργαστήκαμε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αντικειμενική και σωστή και πράγματι πιστεύουμε ότι είναι ο πιο στέρεος τρόπος να ορίσουμε τις ποσοστώσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή στην καταλήψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τη θέση των εμπορικών μας εταίρων στον ΠΟΕ, για παράδειγμα αναφέρατε τη Νέα Ζηλανδία και δεν είναι δεν θα πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες κριτικές όσον αφορά, τη χρήση, όσον αφορά την αύξηση της ε, πρόσβασης ε, στην αγορά της Ευρώπης των 27 συν το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς ε, έχουμε την ξεκάθαρη άποψη ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την πρόσβαση στην αγορά ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Εάν υπάρχει αυτό ε, αυτή τη στιγμή θα είναι και 100 μελλοντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και η πρόταση του, της Νέας Ζηλανδίας κάπως δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά την ε, αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Τελωνιακή Ένωση. Αυτή τη στιγμή εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την Τελωνιακή Ένωση ε, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ε, διαχείριση της ε, κατάστασης. Επίτα υπήρξαν δύο τεχνικές ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσει στο δεύτερο γύρο ο συνάδελφος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, τις, για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε την πρόταση αυτή και θα ήθελα να ολοκληρώσω με το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το ερώτημα του πότε θα εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την Τελωνιακή Ένωση είναι κάπως σαφής, αβέβαιη αυτή τη στιγμή. Και η Επιτροπή στην περίπτωση αυτή είπε Ωραία, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, δηλαδή να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, χωρίς μεταβατική πορεία και χωρίς καμία τελωνιακή συμφωνία και αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ε, 31 Μαρτίου το επόμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή και επειδή η εφαρμογή των χωριστών ποσοστώσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτήσει ορισμένες τεχνικής φύσεως διατάξεις, πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να έχουμε αυτή την πρόταση που, έχουν, θα εγκρίνει οι στο τέλος του χρόνου και θα είμαστε παρκώς προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο στην περίπτωση που τα πράγματα πάνε καλύτερα και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια μεταβατική περίοδο, βέβαια θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό είμαστε προετοιμασμένοι, όπω είπα, για το χειρότερο σενάριο. Με την άδειά σα θα δώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφο για την απάντηση των τεχνικών ερωτήσεων. Καλημέρα σας. Για ρωτήσω για το ερώτημα για το Ρότερνταμ θα πρέπει να επανέλθω στην αρχή αυτή τη μεθοδολογία. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τι ε, διαταράξει στο υπάρχον καθεστώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα καλύτερα δυνατά δεδομένα. Γι' αυτό έχουμε τη μέθοδο του Rotterdam. Ε, το ίδιο βεβαίω συμβαίνει και στο Αμβούργο κλπ. Σαν ε, λύση λοιπόν έχουμε τα εξή. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό, εάν τα δείτε, δεν χρησιμοποιούμε τα συνήθη δεδομένα, γιατί αυτά δεν θα περιλάβουν το Rotterdam Effect. Και θα βαφιστούμε στα δεδομένα που αφορούν τις ε, εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις και όχι το χώρο εισαγωγών. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, υποθέσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να εισαγάγει πουλερικά, θα ζητήσει μια άδεια για να το κάνει. Και αυτή η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να εισαχθεί στο Ρότερνταμ ή στο Αμβούργο. Και αν ε, ο επιχειρηματίας είναι εγκαταστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε είναι υπόλογος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ε, είναι εγκατεστημένο σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα είναι ε, υπόλογο στο εκεί σύστημα. Άρα λοιπόν, και η δεύτερη προσέγγιση είναι εξή. Ε, Είμαστε ανοιχτοί στη Γενέβη για να εξετάσουμε τα βέλτιστα δεδομένα. Αν υπάρξουν καλύτερα δεδομένα, ε, θα τα συμπεριλάβουμε ούτε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις, ε, τα προβλήματα στο εμπόριο. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα βέλτιστα δυνατά δεδομένα που αφορούν ε, την χορήγηση αδειών και θα αναμένουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα δεδομένα που αφορούν τις επιπτώσεις στο εμπόριο. Το δεύτερο ε, ήταν ε, το κομμάτι του TRQ το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και εδώ θα εφαρμόσουμε την εξή μεθοδολογία. Α πούμε ότι είναι 100, τα 50 έχει χρησιμοποιηθεί και το 50 δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Θα δούμε ποιο είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή χρησιμοποίησαν 25 και η Ευρωπαϊκή Ένωση 25. Το 50% εφαρμόζεται στο πλήρες TRQ, δηλαδή στην πράξη έχουμε ένα ποσοστό 50 για το Ηνωμένο Βασίλειο και 50 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν δούμε το κομμάτι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, θα καταλήξουμε στο 25 για το Ηνωμένο Βασίλειο και το υπόλοιπο θα, ε, θα, ε, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Um, then there's one other issue. Επίσης υπήρξε ένα άλλο θέμα ότι ορισμένε φορέ τα TRQs, ποσοστώσει δεν χρησιμοποιούνται καθόλου γιατί εφόσον ε, δεν είναι κατάλληλη κατάσταση τη αγοράς ή γιατί τα, ωφέλη των, ε, δεν, τα οικονομικά ωφέλη δεν είναι τόσο μεγάλα. Εδώ υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε θα δούμε το TRQ του ομοειδούς προϊόντος και θα δούμε το μερίδιο του Ηνωμένου Βασίλειου σε αυτό το TRQ γιατί πρόκειται για ένα πανομοιότυπο προϊόν και αυτό είναι το πιο κοντινό που μπορούμε να πάρουμε ως τα δεδομένα. Δεν υπάρχει τέτοιο TRQ. Εάν, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν υπάρχει πανομοιότυπο, θα δούμε τι γίνεται στο εμπόριο εκτός του TRQ για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Δηλαδή δεν θα παρατηρήσουμε ε, το εμπόριο εντός του TRQ, αλλά εκτός ε, εντός άλλων ε, ε, μοντέλων. Και θα δούμε εδώ πόσο πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πόσο πήγε στις 27 και θα καταλήξουμε και πάλι σε ένα μερίδιο το οποίο θα εφαρμοστεί στο TRQ. Άρα υπάρχει μια συνεπής μεθοδολογία, τη βλέπετε στο παράρτημα για όλα τα TRQ και όπως σας είπα, ο βασικός σκοπός, ο βασικό σκεπτικό ήταν να ελεγχιστοποιηθούν τα προβλήματα στο εμπόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκατε πολύ βαθιά στην μεθοδολογία. Βεβαίω ε, και οι άλλοι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν. Ε, ποια είναι η προσδοκία λοιπόν, θα υπάρξει συμφωνία στον ΠΟΕ ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη κάποιες επαφές με τους εταίρους μας τον ΠΟΕ άτυπες και όπως είπα ήδη δεν έχουμε ομόφωνη στήριξη αλλά για την μεθοδολογία είπαμε στους εμπορικούς μας εταίρους βρείτε μας μια καλύτερη, πιο αντικειμενική μεθοδολογία να την κοιτάξουμε και δεν έχουμε λάβει κάτι. Οπότε η αντίδραση που λάβαμε ήταν περισσότερο πολιτική με την έννοια ότι είπαν θέλουμε να αυξήσουμε την πρόσβαση στην αγορά η ΔΕΟΔΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει η 27 δηλαδή να διατηρήσουν το 100% και το Ηνωμένο Βασίλειο να πάρει κάποιο ποσοστό. Οπότε δεν ξέρω αν θα ξεπερνούσαμε το 100% αλλά έχουμε λάβει κάποιες προτάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό στόχο και μια πιο εύρωστη μεθοδολογία. Για το δεύτερο μέρος της ε, ερώτησής σας, εάν πρέπει να συμφωνήσουν. Εκεί η ανάλυση μας είναι ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή ε, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Γάτ και αυτό θα κάνουμε το επόμενο εξάμεινο αλλά επίσης η ανάλυση μας λέει ότι αν δεν προκύψει συμφωνία έχουμε δικαίωμα σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ να το κάνουμε μονομερός βεβαίως ε, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ακολουθήσουν οι εταίροι μας αλλά και να μας πάνε στο πάνελ. Αλλά έχουμε καλά νομικά επιχειρήματα να πούμε ότι εάν δεν υπάρξει κάτι τότε δικαιούμεθα να το κάνουμε μόνοι μας με, όταν θα αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Τελωνιακή Ένωση. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ακόμα ερωτήσεις. David και Helmut νομίζω είναι μια λογική προσέγγιση υπό τις συνθήκες. Αλλά εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να μείνει στην Τελωνιακή Ένωση, υπάρχει λόγος να σπάσει η ποσόστοση και να την χωρίσουμε. Και μία ακόμα ερώτηση από εμένα. Σε ποιο βαθμό θα υπάρξει κοινή δράση σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την ε, σύμφωνα με την συμφωνία αυτή λοιπόν υπάρχουν ε, Κινέζας ή υπάρχουν ήδη από τώρα διαφορετικές κινήσεις ε, των δύο πλευρών ναι, για την πρώτη ερώτηση υποθετική ερώτηση. Αν έμενε στην ε, Τελωνιακή Ένωση του Ηνωμένου Βασίλειου δεν θα υπήρχε λόγος να χωρίσουν οι ποσοστώσεις. Οπότε πράγματι δεν θα είχε νόημα η προσέγγιση μας. Αλλά εμείς εργαζόμαστε με βάση τις δεδηλωμένες προθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα φύγουν δηλαδή από την Τελωνιακή Ένωση. Δεν είμαι 100% σίγουρος εάν κατάλαβα τώρα την άλλη ερώτησή σας, αλλά εάν έχουμε συμφωνία στη Γενέβη με τους εταίρους του ΠΟΕ. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να κυρωθεί από τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο δηλαδή, με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Και για να προσαρμόσουμε το παράρτημα που έχετε μπροστά σας σε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία στην Γενέβη, έχουμε προβλέψει ε, η Κομισιόν μετά να κάνει τις απαραίτητε τεχνικές προσαρμογές, αλλά και πάλι βεβαίω θα πρέπει να κυρωθεί η συμφωνία από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, κοντελίδε. Α, συγγνώμη. Όσο περισσότερο τα κοιτάει κανείς, τόσο πιο περιπλοκά γίνονται. Έχω μία ερώτηση. Ποια σενάρια εξετάζετε Εργάζεται με βάση το ότι θα φύγει από την Τελωνιακή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά περιλαμβάνεται στην συμφωνία και μια εναλλακτική για την Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε φτιάχνετε και σενάριο με ποσοστώσεις όπου εντός του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν διαφορετικές αναλογίες γιατί και ε, ένα μέρος της, αναλογίας, της ποσόστοσης αφορά την Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, έχουμε μια τεχνική συνάντηση το απόγευμα που θα περίμενα αυτή την ερώτηση. Αλλά πιο σοβαρά τώρα. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση γιατί όπως ξέρετε η λύση αυτή για την Βόρεια Ιρλανδία είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει κάποιο κείμενο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Οπότε κάνουμε μόνο εικασίες. Τότε αυτό το οποίο μπορώ να πω επί της αρχής είναι ότι η κατανομή θα αφορά τους 27 ε, των ποσοστώσεων και για το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν θα είναι ε, μέλος ε, της Τελωνιακής Ένωσης θα ισχύει η ποσόστοση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή είναι η γενική αρχή, αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τι θα γίνει. Οπότε δεν είναι οριστική η απάντησή μου. Μπορεί σε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες να μην ισχύει πια. Ναι, ναι, η ομίχλη είναι έντονη. Λοιπόν, κοντελίβε. Το ωραίο με τους αλγόριθμους ε, είναι ότι μπορεί να αλλάξουν ανα πάση στιγμή οι αριθμοί. Δηλαδή μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο σχήμα απλά ακόμα και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου με συγκεκριμένες περιφερειές και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα οποία συζητάμε, σας είπα, δεν είναι πολύ νομοθετικό έργο, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε πλήρως με το προτινόμενο σχήμα ότι είναι δηλαδή ο σωστός τρόπος για να καταλήξουμε σε ένα πρώτο αποτέλεσμα. Το απόγευμα θα υπάρξει μια τεχνική ενημέρωση και πρέπει να πω ειλικρινά ότι ελπίζω να... ότι Ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε με κάποιες σταθερές ε, συνθήκες για να μην τα αλλάζουμε συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό το Σεπτέμβριο και θα συστήσουμε το σχέδιο έκθεση. Τώρα θα πάμε στο σημείο 9, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων από την ε, τελευταία μας συνάντηση Μέχρι σήμερα έγιναν δύο συναντήσεις στη Νότια Ασία στις 26 Ιουνίου και θα, ακολουθήσουμε τη θα ακούσουμε τη σχετική έκθεση. Κύριε Πράδρε, σας ευχαριστώ. Πράγματι, αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση έλαβε χώρα και μας βοήθησε να τονίσουμε και πάλι το γεγονός ότι η Επιτροπή Ίντα και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων στο Κοινοβούλιο συγκεντρώνεται στις σχέσεις μας με τον Μπαγκλατές αυτή τη στιγμή και θέλουμε να διατηρήσουμε τη θετική μας δέσμευση ούτως ώστε να συνεχίσουν να κινούνται τα πράγματα με έναν επικοδομητικό τρόπο ε, με την ελπίδα περαιτέρω ε, πρόοδων ε, σχέση με τα αποτελέσματα που θα μας έρθουν από τον Μπαγκλαντές. Αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας και πρόκειται για μια σοβαρή δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες και ο Καναδάς. Μέρες, τις μέρες που ακόμα είπα πίστευαν στην αξία του διεθνού εμπορίου. Και ε, η ILO ε, και τη δέσμευση της ε, κυβέρνηση των Μπαγκλατές να βελτιώσει τις ε, συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα του εμπορίου ο αξιότιμος Υπουργός Εμπορίου και ο κ. Χάρπ, ο οποίος είναι Υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές ε, συναντήθηκαν μαζί μας. Ήταν μια σημαντική συνάντηση και ε, τα αποτελέσματα, τα συμπέρασματα ήταν εξή. Το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθάει την ανάπτυξη και την ε, ευημερία στον ε, Μπαγκλαντές. Είναι η δεύτερη εξαγωγική χώρα στο κόσμο. Είναι και το Μπαγκλαντές έχει βασικά ωφέλη. Η EBA έχει μια ξεκάθαρη πρόσβαση στο Μπαγκλαντές και εισφέρει στην ανάπτυξη του Μπαγκλαντές ε, δημιουργώντας ε, πάρα πολλές ε, ευκαιρίες και αυτό το διαπίστωσαν οι υπουργοί του Μπαγκλαντές όπου πολλοί εργαζόμενοι είναι και γυναίκες και αυτό ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα γιατί βλέπουμε ότι αντιμετωπίζονται μέσω του εμπορίου και ζητήματα που αφορούν τη διάσταση του φύλου. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πολύ αξιόλογη πτυχή. Η δεύτερη, η δεύτερη σημαντική δέσμευση αφορά την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ αξιολογήσαμε τις βελτιώσεις ορισμένου τομεί θετικά όσον αφορά την ασφάλεια στον χώρο εργασία, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν δύο θέματα ειδικότερα. Η ευθυγράμμιση με τον εργασιακό νόμο του Μπαγκλαντές ε, σε συμφωνία με την σύμβαση του ILO. Ε, ακούσαμε τους υπουργού ότι έχει θεσπιστεί ένας ε, νόμος, ε, θεσπίστηκε αρχικά, ο οποίος στη συνέχεια όμως αποσύρθηκε και τροποποιήθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μια ανάληψη δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, ίσως το Σεπτέμβριο αυτού του έτους. Αλλά αυτή η χρονική προσταθεσμία θα πρέπει να γίνει σεβαστή και αυτό το τονίσαμε κατά την επίσκεψή μας. Δεύτερον, η συνέχιση της συμφωνίας, γιατί δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα ε, όσον αφορά τις ε, νομικές ε, διενέξεις γύρω από την συμφωνία και θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Και γνωρίζουμε ότι η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου ε, το διαπίστωσε αυτό επίσης σε μια επίσκεψή της ε, στο Μπαγκλαντές. Και εγώ ο ίδιος ε, απέστειλα, ε, θέλω να αποστείλω μια επιτροπή προς τις αρχές του Μπαγκλαντές ζητώντας ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και υπενθυμίζοντάς τους ότι η επιτροπή μας πρόκειται να συνεχίσει να υποθυμίζει στο Μπαγκλαντές τις ευθύνες τους ούτως ώστε να τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, ως ε, συνομοθέτες ε, του κανονισμού έχουμε αυτή την ε, ευθύνη. Και όταν συνταχθεί αυτή η επιστολή θα την κυκλοφορήσω στους συναδέλφους. Επίσης, ασχολήθηκα, συμμετείχα δύο άλλες ενδιαφέρουσες συνδιασκέψεις, μία άλλη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μία άλλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ε, διατύπωσα αυτές τις θέσεις και θα πάω σε μία άλλη συνδιάσκεψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα επαναλάβω αυτή τη θέση. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όταν ε, θέτουμε το ζήτημα αυτό του σεβασμού ε, του χρονοδιαγράμματος θα σφέρουμε θετικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σημαντική δουλειά. Και νομίζω πως είναι καλό που προσφέρουμε μια σταθερή βάση στην κυβέρνηση Βαγκλαντές για τις δεσμεύσεις. Α, κάτι άλλο, στραφούμε τώρα στο Μερκοσούρ. Στις 21 Ιουνίου είχαμε την ε, συνάντηση με το Μερκοσούρ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα που είναι ο εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως είχαμε την ομάδα ε, τη συνεδρίαση της ομάδας μάλλον ε, με τους εκπροσώπους του Μερκοσούρ όπου η επικεφαλής των διαπραγματεύσεων μας εξήγησε τα αποτελέσματα της τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων στην Ουρουγουάη μας ε, μεταβίβασε μια εντύπωση ότι επικρατεί κάποια ανησυχία όσον αφορά αυτόν το γύρο. Εξήγησε πως ορισμένα θέματα ε, που ε, ενδιαφέρον τη διαπραγμάτευση δεν προσεγγίστηκαν στη διάρκεια αυτής ε, της ε, συνεδρίασης. Αμέσως μετά όμως υπήρξαν κάποιες εξελίξεις μετά από την επαφή μεταξύ της Επιτρόπου Μάλστρομ και του Υπουργού της Ουρουάης που προεδρεύει αυτή τη στιγμή στο Μερκοσούρ ε, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται ο γύρος διαπραγματεύσεων. Ελπίζω, υπάρχουν κάποιε ελπίδε να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσει που εξελίσσονται εδώ και πάνω από 20 χρόνια, όπως ξέρετε να ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει μια ετήσια υπουργική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΕΛΑΚ και Εκεί ε, τα μέλη του Μερκοσούρου θεωρούν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους εάν όντως στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας ε, λυθούν τα ευκρεμή θέματα. Το κομμάτι το πολιτικό της συνεργασίας έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τη δική μας διεπροματεύθρια, το 90% των εμπορικών διαπραγματεύσεων έχει επίσης ολοκληρωθεί και μένει ένα 10% το οποίο εστιάζεται βασικά στο περίπλοκο θέμα των αυτοκινήτων, των γεωγραφικών ενδείξεων, όπου ο αριθμός είναι πολύ ψηλός ακόμα. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που πρέπει ακόμα να βγουν για τις θαλάσσιες μεταφορές, την αυσιπλοεία και στο θέμα των αυτοκινήτων έχουμε, ε, έχουμε και κάποια ευαίσθητα προϊόντα ε, του γεωργικού τομέα. Αυτή είναι η κατάσταση. Στη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα σημειωθούν κάποιε πρόοδοι ώστε οι υπουργοί στην τελευταίο γύρο αυτών των ε, υπουργική τη ΕΛΑΚ να μπορέσουν να κλείσουν αυτή την μακρά διαπραγματευτική περίοδο. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κεφαλή των διαπραγματεύσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη λείπουν, ε, χρειάζονται ακόμα δύο εβδομάδες τεχνικών διαπραγματεύσεων, αλλά εφόσον υπάρχει βούληση μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Εγώ είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα γύρο για να κάνω μια σφιγμομέτρηση με τα μέλη του Μερκοσούρ και φαίνεται πως υπάρχει αυτή η βούληση και το πλαίσιο δεν είναι εύκολο. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις ευαισθησίες που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές και νομίζω πως ο στόχος της επίτευξης μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης συμφωνίας ε, ισχύει. Το θέμα είναι αν υπάρχει και η πολιτική βούληση. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. μου του μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συγητή για την ενημέρωση. Δυστυχώς εγώ δεν συμμετείχα, αλλά λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην ε, Βραζιλία με την σχετική νομοθεσία Αναρωτιέμαι αν οι προδιαγραφές που θέτουν οι δύο εταίροι στην συμφωνία θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της ρυθμιστικής ε, προσέγγισης και κάθε δημοκρατικό σώμα έχει δικαίωμα να θέσει προδιαγραφές, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια ξεκάθαρη παραβίαση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που έχουμε εμείς εδώ. με την χρήση ζυζανιοκτών κτλ. Οπότε μπορεί βεβαίως να δημιουργήσει περιπλοκές και ε, το έχουμε συζητήσει τι κάνουμε εμείς εδώ και πώς αντιδράει η Βραζιλία και οι άλλοι εταίροι του Μερκοσούρ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω πως δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για τα θέματα του περιβάλλοντος, γιατί είναι θέματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ξεκάθαρα τη διαπραγματευτική της θέση. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίως στο αν είμαστε πρόθυμοι να κλείσουμε την διαπραγματευτική διαδικασία. Όπως γνωρίζει η συνάδελφος, ε, ο συνάδελφος, εμείς διαπραγματευόμαστε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο όνομα των 28 διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα σημαντικά θέματα έχουν πια επιληθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατηρήσει τις αρμοδιότητές της σε αυτό το θέμα και έχω την εντύπωση πως οι ρυθμίσεις που θα είναι μέσα σε αυτή τη ε, συμφωνία θα πρέπει να τηρήσουν τις διεθνείς, τα διεθνή πρότυπα όπως κάναμε και για την Ιαπωνία, ή τον Καναδά, ε, το Μεξικό πρόσφατα για να μιλήσω και για μια χώρα που βρίσκεται στην ίδια Ήπειρο και εγώ λοιπόν δεν συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες που εξέφρασε <laughs> ο κύριος Σόλτσε Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι αυτή, αυτό το εγχείρημα είναι πολύ ευρύ. Έχουμε, το, είχαμε το χρόνο για να εμβαθύνουμε σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και στα στάνταρα ε, για το κάθε θέμα και νομίζω ότι η ε, Κομισιόν έχει κάνει πολύ επιμελώς τη δουλειά της. Δεν πρέπει αυτό να μας ανησυχήσει λοιπόν τώρα. Το πρόβλημα είναι οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των κανόνων διοδότησης των αυτοκινήτων που είναι ένας επιθετικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το θέμα του κρέατος είναι 99 ε, χιλιάδες ε, τόνοι ε, Ε, είναι, λοιπόν, ε, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την υπόθεση των γεωγραφικών ενδείξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 350 ε, ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης που θέλει να προστατεύσει. Έχει και η Μερκοσούρ 47 ε, και πρέπει και αυτό το νούμερο να διατηρηθεί. Πρέπει να παραμένουμε στα περιθώρια, στα περιθώρια που διατηρήσαμε με τον Καναδά ή με το Μεξικό για να τα τοποθετήσουμε έτσι ώστε να προστατευτούν τα δικά μας σήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να ε, επιτύχει υποχωρήσεις και σε άλλα θέματα όπως την αυσιπλοεία για προϊόντα στο γαλακτοκομικό τομέα και σε αυτά εστιάζονται οι βασικές μας ανησυχίες για την ώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόοδο, πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρότητα με την οποία ε, ε, ε, παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία η Κομισιόν και έχω την εντύπωση, όπως σας έλεγα και στην αρχή, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε αν σε μια τόσο δύσκολη στιγμή μια τέτοιο μεγέθο συμφωνία θα μπορέσει να δώσει ένα μήνυμα σαφούς υπεράσπισης του ελεύθερου εμπορίου και κατά των προστατευτικών τάσεων. Θέλουμε να εξισορροπήσουμε τα, όλα αυτά τα συμφέροντα. Οι εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν κάθε χρόνο πάνω από 4 δι δασμού στις χώρες του Μερκοσούρ και αυτέ είναι οι χώρε οι μόνες τη Λατινική Αμερική που δεν μπορούν να εξάγουν με προτιμησιακό καθεστώ. Πέρα λοιπόν από την οικονομική σημασία, πέρα από την αύξηση του εμπορίου, πέρα από τη σημασία των επενδύσεων, αυτή τη στιγμή διακυβεύεται μια συμφωνία στρατηγική σημασία, όπου οι τεχνικέ ρυθμιστικέ πτυχέ είναι πτυχέ τι οποίε έχει λάβει υπόψη επαρκώ και συζητήσει επαρκώ η Κομισιόν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε με κινητοποίηση τη κοινή γνώμη και τη πολιτική γνώμη, με όλη την ευαισθησία ώστε οι τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που επηρεάζονται να ε, βγουν ωφελημένοι από αυτήν τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες λεπτομέρειες αλλά όντως πιστεύω ότι μια γενική προσπάθεια όσον αφορά ειδικά την αυτοκινητοβιομηχανία, εφόσον έχουμε πρόβλημα με άλλους εμπορικούς μας εταίρους, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείο 10. Λοιπόν, ο εισηγητής ε, για τον γενικό προϋπολογισμό δεν είναι εδώ. Έχουμε όμως την πρότασή του αλλά δεν είναι εδώ και οι σκιώδεις εισηγητές. Ο Κρίστοφερ Χιόλιαν δεν είναι εδώ. Τον αντικαθιστά κανείς. Παρακαλώ. Ε, να μιλήσω εγώ εξ του Κρίστοφερ, αλλά δεν έχω την πρόταση του εισηγητή. Να σας πω τι θα έλεγε ο Κρίστοφερ. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις και ο Κρίστοφερ Φιέλνερ δεν μπόρεσε να έρθει αλλά ε, θέλω να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019 Έχουμε έναν προπολογισμό που θα πρέπει να δώσει αυξημένη χρηματοδότηση για την πιο φιλόδοξη ατζέντα μας μεταξύ αυτών και το μέσο βοήθεια για εμπόριο και βεβαίω αυτό περιλαμβάνει και κονδυλία για την ανάλυση ε, και βεβαίω ε, τους συμμετέχοντες ε, στο Διεθνέ Γραφείο Εργασία. Και το ΕΛΚΑ τονίζει την ανάγκη οι πρωτοβουλίες να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα ωφέλη τη εμπορικής πολιτικής. Όμως, τονίζουμε την ανάγκη η γνωμοδότηση να βασίζεται στον πραγματικό προπολογισμό του 2019 και την σημασία του για την εμπορική πολιτική. Ενώ λοιπόν το Brexit και οι σχετικές συζητήσεις για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικά θέματα για το επόμενο έτος, δεν θα πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ σε αυτήν την γνωμοδότηση. Ο Κρίστοφερ θα υποβάλει τροπολογίες πιθανότατα για την ανάγκη συνοχής της πολιτικής με την εξωτερική πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική την... και τα προγράμματα μακροοικονομικής βοήθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, David Martin για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μας ε, προξενεί εντύπωση το ότι ο εισηγητής υπέβαλε μια λογική πρόταση και υποστηρίζουμε τέσσερις από τις πέντε παραγράφους, δεν υποστηρίζουμε την παράγραφο του Brexit, δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, όπως έχει περιληφθεί εδώ. Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη ουσία τα κεφάλαια που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών κτλ. Οπότε θα υποβάλουμε κάποιες σχετικές ε, τροπολογίες, αλλά ε, κατά λοιπά μας προξενεί και μας έκπληξη. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, γνωμοδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της. Σας ευχαριστώ, Έμα, εξ ονόματος του κυρίου Λούνες, μα κανείς δεν είναι εδώ σήμερα. Το ECR θέλει ο προπολογισμό αυτός να στοχεύει την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία, της νέες προκλήσεις και βεβαίως να έχουμε αναδιάταξη αντί για νέα κονδύλια. Γι' αυτό ψηφίσαμε κατά της εντολής για μετά τον τριμερή διάλογο και αυτό το οποίο μας ανησυχεί περισσότερο ε, είναι ακριβώς παραγραφός 4 που προτείνει ή ΜΚΟ που είναι κατά του ελευθέρου εμπορίου να χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό βιολογισμό. Είμαστε κατά αυτής της σπατάλης δημοσίου χρήματος. Σας ευχαριστώ. Μαρίτια Χάκε δεν είναι εδώ, Χάιντι Χάουταλα δεν είναι εδώ, Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ επίσης να πω ότι σε γενικές γραμμές πηγαίνει σε μια σωστή θα έλεγα κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θέλω να παρατηρήσω ότι Μάλλον πρέπει να τονίσουμε περισσότερο κάποιες νέες πτυχές της στρατηγικής εμπόριο για όλους που ε, ακολουθεί αυτή η Κομισιόν για να ενταχθεί και στον προπολογισμό του 2019 να τονίσουμε τα ζητήματα δίκαιου εμπορίου που πρέπει να αναφερθούν. Επίσης συμφωνώ ότι οι μικρόμεσες επιχειρήσεις είναι κάτι το σημαντικό και τέταρτον θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες προσθήκες ε, στο σχέδιο πρότασης ε, που θα αφορούν την εφαρμογή του κενικευμένου συστήματος προτιμήσεων, όπως επίσης και κάποιες πτυχές ε, κάποιων διμερών συμφωνιών που πρέπει να συνοδεύσουν την διαδικασία αυτή του follow-up, ειδικά στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπου μόλις φέτος ε, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κομισιόν. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ε, η Κομισιόν θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι ο προϋπολογισμός του 19 καλύπτει τις ανάγκες μας. Έχουμε έναν μικρό λειτουργικό προϋπολογισμό και επίσης χρησιμοποιούμε και τα μέσα που υπάρχουν ε, στον προϋπολογισμό εξωτερικής ε, δράσης ε, και τα περισσότερα ζητήματα που αναφέρατε στις παρεμβάσεις σας καλύπτονται είτε από τον λειτουργικό προϋπολογισμό είτε από τα εξωτερικά μέσα έχουμε χρησιμοποιήσει και πάλι τον πολύ μικρό προϋπολογισμό μας για να αξιολογήσουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες, για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις ε, διαπραγματεύσεις και στον μηχανισμό εφαρμογής. Επίσης ε, χρησιμοποιούμε ένα από τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής ε, για να χρηματοδοτήσουμε έργα και θεωρούμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμούς έχει για του χρόνου θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τις ε, προτεραιότητές μας ε, όπως έγινε και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς και στον τομέα βοήθεια έναντι εμπορίου και πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό αυτόν για να προωθούμε και ζητήματα δικαίου εμπορίου όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια και επίσης ε, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα έργο το οποίο εφαρμόζαμε ήδη φέτος ε, και ίσως τελικά συνεχίσουμε με τον προπολογισμό του 2019 με τον δικό μας λειτουργικό προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορεί να ολοκληρώσει ο εισήγητης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ το ότι δώσατε τον λόγο πρώτα στους σκιώδεις εισηγητές. Πολύ επικοδομητικό πραγματικά προεδρεύεται εξαιρετικά. Είναι πολύ σύντομη αυτή η γνωμοδότηση εν μέρη γιατί ε, πολλά από αυτά τα οποία έβαλα τα κόψαν οι συνάδελφοι και εγώ κόψα πολλά από αυτά τα οποία έβαλαν οι συνάδελφοι. Αλλά ως έχει δεν ξέρω εάν θα αλλάξει πλέον σε ένα θεσμικό όργανο που υπάρχουν πάρα πολλά μακροσκελή πράγματα ίσως αξίζει που και που να έχουμε κανένα κείμενο το οποίο θα είναι συνοπτικό. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Οπωσδήποτε θα ψηφιστεί και θα δούμε μετά εάν θα μπορέσω να στηρίξω την γνωμοδότηση μετά από τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο το διαχειριστήκατε. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάρτμος. Πράγματι υπάρχει δυνατότητα υποβολής ε, τροπολογιών μέχρι τις 13 Ιουλίου στις 12 η ώρα. Και στις 20 Ιουλίου 6 ώρα μέχρι τις 20 Ιουλίου 6 ώρα για τις ε, τροπολογίες του προπολογισμού. Η πρώτη είναι μεσημέρι και η άλλη είναι 6 απόγευμα. Και θα εγκρίνουμε την σύσταση του κυρίου Ντάτμουθ ε, για τις 29 Αυγούστου. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 11 το blockchain την τεχνολογία αυτήν και τις συνέπειες που έχει στην εμπορική πολιτική. Η συγγήτρια είναι η Εύα Μακλάρκιν, στην οποία δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε το blockchain και το τι σημαίνει για το διεθνές εμπόριο. Πολύ συναρπαστικό θέμα θα έχετε δει τις εκδηλώσεις ε, που γίνονται και νομίζω ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι πλέον ε, το αντιλαμβάνονται και αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να δούμε τις ε, σχετικές τεχνολογίες για σκοπούς διεθνούς εμπορίου. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να υπάρξει μια επανάσταση στο εμπόριο και στην ανταλλαγή αγαθών και ιδεών. Και πριν περάσω σε αυτό θα ήθελα να, κάνω κάποια σχόλια για την τεχνολογία. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε το πώς λειτουργεί. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν επιτρέπει σε διαφορετικά μέρη να κάνουν ασφαλείς συναλλαγές χωρίς την ανάγκη κάποιου ενδιάμεσο. Κάποια από αυτά είναι μια τεχνολογία διανεμημένων βάσεων δεδομένων όπου καταχωρούνται άπαξ οι συναλλαγές και δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν. Τις λέμε διανεμημένες γιατί υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα του συστήματος ε, που αναβαθμίζονται με βάση έναν συνενετικό αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ποιο μπλοκ θα προσθεθεί στην ναι. αλυσίδα. Λοιπόν, ελπίζω να καταλαβαίνετε ακόμα να παρακολουθείτε. Λοιπόν, όχι. Οπότε έχουμε σε κάθε φορά μία προσθήκη ε, ενός μπλοκ που προστίθεται με ένα χάσμα υπογραφή θα λέγαμε και υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ε, blockchain. Υπάρχουν όπως είπαμε οι βάσεις δεδομένων ή δημόσιες και ιδιωτικές. Τις δημόσιες μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει και να συμμετέχει στον αλγόριθμο όπως το bitcoin, το ethereum και τα άλλα κρυπτονομίσματα. Να σας πω λοιπόν ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτόν τον τύπο βάσεων δεδομένων. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για την ασφάλεια και τη χρησιμότητα αυτής της τεχνολογίας. Αντιθέτως η έκθεσή μου θα εστιαστεί στις, ε, στα blockchain ιδιωτικής άδειας ε, που μοιάζουν ε, με μια παραδοσιακή βάση δεδομένων όπου επιλέγονται οι χρήστες. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται εκεί δεν μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν και τα διαχειρίζονται οι διαχειριστές του δικτύου. Οπότε το επίπεδο της ασφάλειας ε, και της εμπιστοσύνης των χρηστών στο ότι δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα εξαρτάται από τους κανόνες που εφαρμόζονται. Και έχουμε άρα ένα επιπλέον στοιχείο ελέγχου των χρηστών και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα την εφαρμογή του στο διεθνές εμπόριο. Είναι λοιπόν ένα θέμα ασφάλειας, διαφάνειας και εμπιστοσύνη στο σύστημα. Γνωρίζω πως κάποιοι βουλευτές ερώτησαν γιατί η Επιτροπή μας πρέπει να ασχοληθεί με την εφαρμογή του blockchain στο διεθνές εμπόριο και γνωρίζω ε, την ανησυχία που εξέφρασαν κάποιοι ότι το blockchain δεν είναι μια μαγική λύση. Ε, πρέπει λοιπόν ακριβώς ε, να μην δημιουργούμε προβλήματα μόνο και μόνο για να τα λύσει το blockchain. Πρέπει ακριβώς να βρούμε μια πιο μετρημένη λύση και να το εκμεταλλευτούμε εκεί όπου προσθέτει κάποια αξία και να μην το χρησιμοποιούμε όταν δεν προσθέτει κάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να εφαρμόσουμε το blockchain στο διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί τομεί στους οποίου μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Μπορεί επίση να μειώσει τα εμπόδια και τους φραγμούς ε, και να προωθήσει το παγκόσμιο εμπόριο κατά 50%, να μειώσει το κόστος ε, των συναλλαγών ε, με το να μην υπάρχουν να μην υπάρχει γραφειοκρατία, να ενισχύσει την ροή δεδομένων για να καταπολεμηθούν τα πλαστά έγγραφα και αγαθά και να βελτιώσει την διαφάνεια ενισχύοντας έτσι την βεβαιότητα για την προέλευση των αγαθών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά πιλωτικά εμπορικά έργα που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος μεταφοράς και να κάνουν ε, την βιομηχανία πιο φιλική προς το περιβάλλον. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα μπορούσαν να ωφεληθούν ε, πολύ από το blockchain. Θα γίνουν πιο εύκολα να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες, με τις αρχές και να μπορέσουν έτσι να αναπτυχθούν. Και όχι μόνο μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι καταναλωτές, που θα έχουν την δυνατότητα να βάλουν κάποια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και να λάβουν άμεσα μία επιβεβαίωση. Επίσης μπορεί να υποστηρίξει το δίκαιο εμπόριο, καθώς τα βιώσιμα αγαθά θα έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την προέλευση, την νομιμότητα ενός προϊόντος, την επεξεργασία του και να μην ε, αγοράζουμε αγαθά από πολέμους, ε, συγκρούσεις ή που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ακριβώς ε, θα μπορούσαμε έτσι, παραδείγματος χάρη συχνά μιλάμε για την χαμηλή χρήση των συμφωνιών ελευθέριου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι περίπλοκοι οι κανόνες για προτιμησιακή πρόσβαση θα μπορούσε το blockchain να απλοποιήσει κατά πολύ τους κανόνες αυτούς και να προωθήσει τις εξαγωγές και υπάρχει δυνατότητα να το εκμεταλλευτούμε στις ε, πολιτικές ε, άμυνας ε, του εμπορίου όταν έχουμε δηλαδή μια πλημμυρίδα προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας το σύστημα γενικεμένων προτιμήσεων. Επίσης μπορεί να εξυγχρονίσει τον σχεδιασμό και την κατανομή των ποσοστώσεων, καθώς θα μπορούσαν έτσι να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά οι τελωνιακές αρχές για να δουν την ζήτηση, την απόδοση και άλλους δείκτες. Ε, θα μπορούσαν έτσι οι τελωνιακές αρχές να αποκτούν αυτομάτως τα απαραίτητα στοιχεία για μια τελωνιακή δήλωση και να μην υπάρχει ανάγκη μιας ε, φυσικής ε, επαλήθευσης των εγγράφων για τα αγαθά που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας έτσι μια διαχείριση κινδύνου και χρησιμοποιώντας ε, τα δεδομένα που υπάρχουν και την ανάγκη για δαπανηρές ε, για να πανηρούς ελέγχους. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι από την φύση και την αρχιτεκτονική του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προστασία των καταναλωτών χωρίς να εμποδιστεί η εξέλιξη του blockchain, κάτι το οποίο βεβαίως είναι δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα με διαλειτουργικότητα έτσι ώστε και οι δημόσιοι φορείς να εκμεταλλευτούν τα θετικά του συστήματος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για νέες εταιρείε που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ψηφιακέ εφαρμογές. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και θα τα γράψω στην έκθεσή μου. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω το εξή ο Τόμας Φρίτμαν είπε ότι ο κόσμος είναι επίπεδος και οι τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα το καθιστούν ακόμα πιο επίπεδο. Και πιστεύω ότι το blockchain είναι η ευκαιρία να επαναστατικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το εμπόριο και οι συναλλαγές και η μείωση των φραγμών κινούνται, εξελίσσονται ταχύτερα. Ε, πρόκειται για μια ορθολογική χρήση της τεχνολογίας, ε, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη παραμένει σε πρωτοπόρα όσον αφορά την χρήση αυτής της τεχνολογίας και θα πρέπει να λάβουμε, πάρουμε δικές μας πρωτοβολίες όλο και συχνότερα. Ε, θα ήθελα να συνεργαστώ με τους συναδέλφους ε, Ούτε ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της ε, τεχνολογίας ε, εχμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε κάθε νέα επανάσταση θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να θεσπιστεί σε σχέση με αυτή την επανάσταση η εκ μέρους του ΕΛΚΕ. Ο συνάδελφος Ανδρικένα είναι ασθενή, δεν μπορεί να παραστεί εδώ και ευχόμαστε καλή... Ε, Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και ο Λανάντου Κένε πιστεύει ότι, είναι μια... ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται στον κατάλληλο χρόνο και θα πρέπει να εξοπλίσουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής, της ε, βράχη και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το διεθνές εμπόριο. Κάτι το οποίο είναι πολύ το φυσιολογικό, εφόσον είμαστε Επιτροπή Εμπορίου. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της κανονιστικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξ αρχής το blockchain έτυχε μεγάλης προσοχής σαν μια πλατφόρμα κρυπτοσυναλλαγών, αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ωστόσο, επειδή είναι νέα τεχνολογία, είναι δύσκολο να ορίσουμε τα όρια και το φάσμα των ευκαιριών που μας ε, παρέχει. Για το διεθνές εμπόριο, το blockchain παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και μπορεί να μας εγγυηθεί ένα ασφαλές και τυποποιημένο εμπόριο χρησιμοποιείται ήδη στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό ε, τομέα καθώς και στον τομέα των μεταφορών και επιτρέπει σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να διευρύνουν τις ευκαιρίες διεθνούς εμπορίου και να βελτιστιοποιήσουν το, τη σχέση κόστους ε, πρόσθετα, το blockchain στηρίζεται στη διεύρυνση του όγκου ε, συναλλαγών. Ε, βεβαίως υπάρχει ένας ε, κίνδυνος απάτης. Τα τελευταία χρόνια τα τρομοκρατικά πλήγματα και οι μεταναστευτικές ροές οδήγησε σε μια αυστηροποίηση των ελέγχων και Ε, με τον τρόπο αυτό ε, υπάρχουν αρνητικές, ε, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και για τις εμπορικές συναλλαγές λόγω των αυστηρών ελέγχων στα σύνορα. Γι' αυτό τράπεζες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο ψάχνουν τρόπους να μειώσουν το κόστος και να επισπεύσουν τις ε, συναλλαγές. Το blockchain είναι μια τέτοια τεχνολογία που επιτρέπει την ε, ε, μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση εμπιστοσύνης σε εμπορικές συναλλαγές και οι εμπορικοί εταίροι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα, τους εμπορικούς όρους. Ε, θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν και ξεκάθαρες κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, μελλοντικά σχέση με αυτή τη νέα μέθοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ε, γκρίζες ζώνες και ερωτηματικά. Η έκθεση αυτή βεβαίως παρουσιάζει τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η νέα τεχνολογία. Το blockchain είναι βρίσκεται στη φάση εισαγωγής και θα πρέπει βεβαίως να αποφύγουμε τις υπερβολικές ε, ρυθμίσεις στην εφαρμογή. Ε, εν κατακλείδη, ε, το blockchain μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση εμπιστοσύνης, ε, δίδοντας, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων, αλλά οι κανόνες προστασίας θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Και αν μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση, Ελπίζω ότι αυτό το, αυτή η μέθοδος πραγματικά ε, ε, θα εφαρμοστεί στην πράξη, παρόλο που εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια σημαντική μέθοδος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική και θα πρέπει να είναι φιλική προς τις καινοτομίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε ενδεχόμενες εφαρμογέ τη μεθοδολογία blockchain. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το πώς μπορεί να δουλέψει η τεχνολογία αυτή, αυξάνοντας τις, πιθαν... Ε, ευκαιρίες για επιχειρηματίες και καταναλωτές και δίνοντας μια δυνατότητα ανείχνευσης των, ε, της Η τεχνολογία αυτή μπορεί να ευεργετήσει επίσης και τις επιχειρήσεις και να δώσει δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν καλύτερα. Επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών και των πολιτών να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αγοράζουν δεν προέρχονται από περιοχές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε το πώς η τεχνολογία blockchain θα μπορέσει να είναι χρήσιμη για τις ε, επιχειρήσεις και να αποτελέσει ένα εργαλείο βιωσιμότητας. Ε, Βεβαίω υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, όπως ήδη υπόθηκε, και θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν. Αλλά εγώ αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία με την συγγέτρια και τους σκιώδεις. Γιατί το έργο μας ως πολιτική είναι να ακούσουμε αυτούς ε, που έχουν γνώση τεχνολογίες και να περάσουμε τις γνώσεις αυτές από ένα πολιτικό φίλτρο. Αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εκπρόσωπος του ΑΛΔΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, Έμα, για τα όσα μας είπε. Μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα για το δυναμικό αυτής της μεθοδολογίας και τα ωφέλη για τη δική μας Επιτροπή. Και έχω εμπιστοσύνη ότι από κοινού ε, θα εκπονήσουμε μια καινοτόμο έκθεση. Αν δούμε τι γίνεται για τα... Ε, βεβαίως, για τα, με τα πνευματικά δικαιώματα ε, θα έπρεπε να είχαμε μια άλλη έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έρχεται τον κατάλληλο χρόνο. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα αυτή τη μεθοδονέα τεχνολογία. Για μα είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε το θέμα ανοιχτόμυαλα, να δούμε πού βρίσκονται ευκαιρίε, πού βρίσκονται ε, δυνητικοί κίνδυνοι, πού θα πρέπει να παρέμβουμε νομοθετικά κλπ. κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, για όλα τα μέρη. Η μεθοδολογία αυτή είναι πολύ χρήσιμη ε, όσον αφορά τους καταναλωτές για σχέση με την προέλευση των προϊόντων, αλλά και για τους επιχειρηματίες σε σχέση με την μείωση του κόστος, ε, επίσης για την ελάφρυνση των δασμολογικών διαδικασιών κλπ ε, επίσης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ε, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και περισσότερη ασφάλεια στις συναλλαγές. Το blockchain έχει το δυναμικό να κινητοποιήσει το ελεύθερο εμπόριο και να οδηγήσει στην ανάκαμψή του και νομίζω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς ε, ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία ε, υπάρχει ένα δυναμικό για το ελεύθερο εμπόριο και το blockchain είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει εδώ. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια θέματα σχέση με τα ιδιωτικά δίκτυα, παραδείγματι, και, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο τι γίνεται στο δημόσιο χώρο, τι είδους ε, προδιαγραφές θα πρέπει να ε, οριστούν εδώ. Ε, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αντικαταστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ποιος θα πρέπει να είναι ο βαθμός διαφάνειας κλπ. Αλλά επίσης να υπάρξει ένας κοινό ορισμός ασφάλειας και αυτό είναι ένα διακύβευμα εδώ και γι' αυτό χαίρομαι για την ε, συνεργασία με την συγκέντρια και τους σκιώδεις, ούτως ώστε να έχουμε πραγματικά μία καινοτόμα έκθεση από την οποία όλοι να υποφεληθούμε. Ευχαριστούμε πολύ ο Κλάους Μπούχνερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ για τα ε, πλεονεκτήματα. Έχουμε ήδη ενημερωθεί από την εισηγήτρια. Νομίζω ότι μας το ανέπτυξε πολύ γλαφυρά. Αλλά όπως και κάθε νέα τεχνολογία, το blockchain συνδέεται με κάποια προβλήματα ένα κομμάτι από αυτά ήδη αναφέρθηκε, θα το πω με τα δικά μου λόγια. Η αποθήκευση η ίδια είναι ασφαλής, γιατί εάν τα δεδομένα καταναμμένα σε χιλιάδες υπολογιστές είναι δύσκολο να υπάρξει χειραγώγηση των δεδομένων. Το πρόβλημα είναι όσον αφορά την εισαγωγή των δεδομένων και στην επιλογή. Και εδώ χρειαζόμαστε ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο ίσως δεν είναι δικό μας καθήκον, αλλά μπορούμε ίσως να συμβάλλουμε εδώ. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω την επόμενη παρατήρηση που υπονοήθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι συγκεχημένα τα όρια μεταξύ ιδιωτικών δεδομένων, ιδιωτικών συσκευών και εμπορίου. Ε, αυτό το οποίο ονομάζουμε πέμπτη γενεά στο διαδίκτυο. Εδώ βεβαίως υπάρχει μια ευκαιρία για τεχνολογία blockchain, χωρίς αυτήν ε, δεν γίνεται προχώρηση στα πράγματα, αλλά από την άλλη εγκυμονούνται μεγάλη κίνδυνο όσον αφορά την προστασία δεδομένων, καθώς και την χειραγώγηση των ε, δεδομένων που εισέρχονται και εξέρχονται. Ε, Υπάρχει ανάγκη λοιπόν μεγαλύτερη ασφάλεια εδώ και θα πρέπει εμεί ε, ε, εδώ, η δική μα επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα αυτό τη προστασία για την είσοδο και την έξοδο των δεδομένων και ελπίζω να είμαστε εδώ αρκετά αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, άκουσα την εισαγωγή της ε, κυρίας ε, Μακλάρκιν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση και χαίρομαι ιδιαίτερος με την ε, σημασία που αποδίδει η κυρία Μακλάρκιν στο blockchain και στην διαφάνεια. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Ποιος ελέγχει την ισχύ των πληροφοριών που αποθηκεύονται. Μπορούμε να ελέγξουμε την προέλευση ενός προϊόντος, αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος εισάγει τις πληροφορίες. Και λέτε πως ε, υπάρχει ο κίνδυνος για να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα το blockchain. Βλέπετε κι εσείς αυτόν τον κίνδυνο. Επίση ε, τι γίνεται όταν υπάρχουν άνισα εμπορικά μπλοκ με διαφορετικές προδιαγραφές. Εν ολίγηση υπάρχουν πράγματι κάποιες ευκαιρίες αλλά και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και αναμένουμε με περιέργεια την περαιτέρω διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με την όχι τόσο αισιόδοξη προσέγγιση των συναδέλφων. Υπάρχουν πράγματι ευκαιρίες και δυνατότητες αλλά μιλάμε για τον τομέα του διεθνούς εμπορίου που σχετίζεται με προϊόντα ή υπηρεσίες. Οπότε το ερώτημα είναι που είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία για το εμπόριο τρίτων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού βρίσκονται οι ε, σερβερ οι οποίοι χρησιμοποιούν τεράστια ενέργεια. Αυτό σημαίνει Και το ε, ερώτημα επίσης είναι πώς γίνεται ακριβώς πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και ποιος συμμετέχει σε αυτή την διάχυση της πληροφορίας. Δεύτερο ερώτημα, σε ποιο βαθμό η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών θα έχει κάποια επίδραση στο πολυμερές εμπορικό σύστημα και στον ΠΟΕ ο ΠΟΕ είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Είμαστε ήδη στο σημείο στο οποίο μπορούμε πραγματικά να πείσουμε και τους εταίρους μας για κάποιες κοινέ προδιαγραφές, τους εταίρους στα πολυμερή φόρουμ. Τρίτον, συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι Πράγματι, κάποια πράγματα φαίνονται αυτή τη στιγμή εφικτά στην ιδιωτική σφαίρα. Το θέμα είναι πώς συνδέονται με, τα, με την δημόσια πτυχή την οποία αναφέρατε και τι θα γίνει με τις εξελίξεις ε, όσον αφορά την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς αυτό. Και η τέταρτη ερώτηση ποιο βαθμό υπάρχει κάποια διαφάνεια των οικονομικών ροών σε αυτό το σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι ε, όταν έχουμε εμπορικές συνομιλίες με τρίτες χώρες, ειδικά στη Λατινική και Νότια Αμερική, ότι υπάρχει πρόσβαση της μαφίας των ναρκωτικών σε διάφορα λεφτά, προϊόντα εγκλήματος ε, που αναζητούν ε, τρόπους να τα αποθηκεύσουν. Ε, μήπως το blockchain είναι ένα ιδεώδες μέσο μέσω της περισσότερης διαφάνειας να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα ή μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ένα επιπρόσθετο στοιχείο ξεπλήματος ε, χρήματος σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην Κομισιόν. Ο κ. Τόμας Μπέρτ, ε, ο τμήματάρχης για την εμπορική στρατηγική. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε και εμείς την ευκαιρία να ακούσουμε και να μάθουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. και ακριβώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στο εμπόριο όσον αφορά τις κανόνες προέλευσης, τις εφοδιαστικές αλυσίδες κτλ. Οπότε μένουμε την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Να επανέλθω λίγο στο ζήτημα. Υπάρχει κάποια σκέψη εντός της Κομισιόν περί blockchain και εμπορίου για τις ε, δυνατότητες και τη σκοτεινή πλευρά της υπόθεσης αυτής ή ε, μαθαίνετε απλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω κάποια θέση της Κομισιόν να αναφέρω σήμερα και να τονίσω ότι και εμείς βλέπουμε πολλές δυνατότητες. Έχουμε διάφορα έργα όχι μόνο στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και στην Γενική Διεύθυνση Ταξούντ και Connect. Βλέπουμε λοιπόν τις δυνατότητες που υπάρχουν και κάποια ρυθμιστικά ζητήματα πράγματι και άρα δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε λοιπόν την συζήτηση στην οποία βεβαίω ε, θα λάβουμε και εμείς μέρος. Ωραιότατα. Έμα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι προφανές ε, γιατί ακριβώς αυτή η Επιτροπή ηγείται ε, με αυτή την έκθεση για το blockchain και έτσι θα μπορέσει και η Κομισιόν να μάθει για αυτή τη τόσο νέα τεχνολογία που ε, ε, αλλάζει ρηξικέλευτα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι υπάρχουν συν και πλήν θετικά και αρνητικά ευκαιρίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και παγίδες που πρέπει να τις κατανοήσουμε καλά. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως την τεχνολογία πώς ε, εφαρμόζεται πριν προχωρήσουμε σε νομοθεσία. Γι' αυτό και πέρασα και ώρα ε, ε, εξηγώντα τι ακριβώς κάνει και πώς λειτουργεί. Γιατί συχνά βοτάμε με τα μούτρα χωρίς να έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί να επανέλθω στο Χιάλμοτεφ, βεβαίω ε, και πιστεύω πως θα πρέπει να βρούμε λύση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του ξεπλήματο χρήματο και όλα αυτά τα θέματα. Φυσικά και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και αυτή η νέα η τεχνολογία με τόσο ασφαλή και διαφανή μητρώα των δεδομένων θα βοηθήσει. Όπως είπα, δεν είναι και το μαγικό ραβδί, ε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Άλλες χώρες ολόκληρο τον κόσμο να πτήσουν αυτή την τεχνολογία και θα τη χρησιμοποιήσουν. Και εμείς πρέπει να έχουμε πάντοτε το πλεονέκτημα, να ηγούμεθα στην ανάπτυξη και κατανόηση αυτής της τεχνολογίας. Γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στο θέμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους ε, σκιώδεις συζητητές και να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να καταλάβει πώς θα μπορέσει να ε, χαλιναγωγήσει αυτή την τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ετοιμαστεί λοιπόν αυτή η έκθεση στη διάρκεια των θερινών διακοπών και θα τη συζητήσουμε στις 29 Αυγούστου. Oh, that may changed. Is my understanding on that date? Ε, νομίζω ίσως αυτό αλλάξει, αλλά θα σας ε, ξανα ε, όταν θα έχει τελειώσει η δουλειά μου. Μάλιστα, θα συζητήσουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο την έκθεση. Μάλιστα, και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών, γιατί περιμένουμε τον Υπουργό ψηφιακών και οικονομικών υποθέσεων και τον την είπα το ε, ε, ε, εκπρόσωπο για το εμπόριο Μαργαρέτα Σάμρογκ. Ευχαριστώ.

Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Χαίρομαι που ήρθε εδώ η Μαργαρέτε Σραμπερκ, συγγνώμη, ομοσπονδιακή υπουργό ψηφιακών και οικονομικών υποθέσεων από την Αυστρία και η οποία είναι αρμόδια για την ε, εμπορική πολιτική και θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. Βεβαίως, εδώ, κύριε Υπουργέ, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε δύο νομοθετήματα τα οποία μας απασχολούν. Ο κύριος Προύς... Ε, um και το δεύτερο νομοθέτημα αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών για προϊόντα τα οποία είναι χρήσιμα τόσο στρατιωτικό όσο και πολιτικό τομέα. Και επίσης το ζήτημα των τεχνολογιών πληροφορίας και εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και μάλιστα ε, σε σχέση για παράδειγμα με τις ε, φήμες ότι η παρακολούθηση της αντιπολίτευσης στην ε, Τουρκία γίνεται με ευρωπαϊκό software. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας μιλήσετε για αυτά. Επίσης τα θέματα που αφορούν την ε, Ιαπωνία και έχει αναβληθεί λόγω της ε, πλημμύρας των ε, καταστροφών στην Ιαπωνία έχει αναβληθεί η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας και, ε, και στα μέσα Οκτωβρίου έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη και ίσως θα γίνει και εκείνη και η υπογραφή της συμφωνίας με την Ιαπωνία την ίδια στιγμή. Είναι δύο σημαντικότατες εμπορικές συμφωνίες. Βεβαίως ε, όλα αυτά σχετίζονται με την εξέλιξη του και την αναδιοργάνωση του παγκοσμίου εμπορικού συστήματος ε, λόγω ακριβώς ε, των προβλημάτων που συνδέονται με τη στάση των ΙΠΑ. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις καθώς και το μέλλον του πολυμερούς συστήματος. Άρα πραγματικά είναι δύσκολη καιρή, κυρία Πρόεδρε, και περιμένουμε με ανησία να μας παρουσιάσετε πώς το, το πώς το αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Για πρώτη φορά έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σήμερα έχω διάφορες ε, συναντήσεις ε, που με ενδιαφέρουν πολύ. Σε σχέση ε, με το τριμερή διάλογο, το FTI screening είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Θα παρίσταμε και θα δω ποιες είναι οι τοποθετήσεις. Ε, κύριε Πρόεδρε, είπατε ήδη, ε, αν τα προβλήματα με τις ε, ΙΠΑ, Βεβαίω οι εξελίξει εδώ δεν είναι καθόλου ικανοποιητικέ. Είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουδέποτε μέχρι τώρα έχει συμφωνήσει με κάτι τέτοιο. Και ε, από κοινού ε, έχουμε μια ισχυρή αγορά με ισχυρέ εξαγωγές και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην κατάσταση της Αυστρίας. Η Αυστρία είναι μια μικρή οικονομία όπου κάθε δεύτερη θέση εργασίας συναρτάται με το εμπόριο και 6 από 10 ευρώ του ΑΕΠ αντιπροσωπεύονται εδώ. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα υποστηρίξουμε στο μέτρο του δυνατό την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει, ούτως ώστε να κατευναστούν οι αγορές. Ο στόχος μας είναι να έχουμε λιγότερους δασμούς, όχι αύξηση των εμπορικών εμπορίων και των δασμών. Ε, ως κάθερο μήνυμα, εμείς σαν Αυστρία πριν από μερικές ε, μέρες επικυρώσαμε τη ΣΕΤΑ ως 12η χώρα. Ε, πριν από εμά ήταν η χωρα πριν απο εμα ηταν η φιλανδια και πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα πρέπει να υπάρξει μια καλή συνεργασία προκειμένου να προωθηθούν τα θέματα τα οποία έχουν τύχει πολύ καλή ε, επεξεργασία και η ΣΕΤΑ είναι μια πολύ καλή εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό θα μεριμνήσουμε ούτε ώστε να εφαρμοστεί αντιστοιχά στι διάφορε ε, χώρε. Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία, Γιατί εμεί ω Προεδρία του Συμβουλίου είμαστε υπό το έμβλημα μια Ευρώπη η οποία προστατεύει, παρέχει προστασία. Και δικό μα μέλημα είναι το θέμα του εμπορίου, μέσω του εμπορίου να αυξηθεί η ευημερία, θέσει απασχόληση επίσης οικονομική μεγέθυνση ε, και όχι να παρεύουμε σε μια φάση όπου τα πράγματα πάνε καλά. Το δικό μας μέλημα είναι να ε, εκπροσωπήσουμε το καλύτερο δυνατό τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες ε, προϋποθέσεις και το καλύτερο πλαίσιο. Γι' αυτό χαίρομαι που διάφοροι οικονομικοί εταίροι, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ και έχουν και, τα πρώτα βήματα προς Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία ε, είχαν μεγάλη υποστήριξη από τη δική μας πλευρά. Τώρα, θα πω στο θέμα FDI screening. Είναι πολύ σημαντικό να εξορροπήσουμε εδώ τα διάφορα αντικρώμενα συμφέροντα ε, και χαίρομαι που θα συζητήσουμε, θα συζητήσω και μαζί σας αυτό το θέμα. Ο στόχος μας είναι κατά τη διάρκεια της θητείας μας να υποστηρίξουμε εντόνως αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ε, καινοτόμες πολυμερείς προσεγγίσεις θα είναι μελλοντικά αναγκαίες. Επίσης το να, ξανα, ε, να επανεξετάσουμε κάποια θέματα, να υποστηρίξουμε και τον ΠΟΕ, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια καινοτόμα διαδικασία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του πολυμερούς ε, συστήματος. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει μια στενή συνεργασία και εντατική συνεργασία και εδώ ήδη έκανα τα πρώτα βήματα τόσο με εσά όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον ίδιο τον ΠΟΕ. Η Σεσίλια Μάλστρομ, η Επίτροπος, έχει την πλήρη μας υποστήριξη και εκείνη βεβαίως έδωσε κάποιες ενδείξεις ε, λέγοντας ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ισχύον σύστημα και να μετεξελιχθεί ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα διάφορα θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Και εδώ είναι σημαντικό να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινηθούμε προς τα μπρος. Χαίρομαι για μια επικοδοματική συνεργασία τους προσεχείς ε, μήνες για την ανταλλαγή απόψεων και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω μια εμπειρία 22 ετών όσον αφορά τη διεύθυνση επιχειρήσεων και ο στόχος μου είναι ε, να προχωρήσουμε σε όσο δυνατόν ε, περισσότερες εφαρμογές συνδέοντας το με ε, ταχύτητα, με τον παράγον ταχύτης και αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, εκπροσώπους της, ε, των ε, Ε, των, ε, ευρωπαϊκών ομάδων, καταρχήν εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Ε, βεβαίως υπάρχει Υπάρχει μια σειρά γενικά, γενικών ε, θεμάτων στην ε, πολιτική εμπορίου, στα οποία αναφερθήκατε. Ε, βεβαίως, πολύ γενικόλογα, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Έχετε μια ιδέα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο ΠΟΕ γιατί ε, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνεται θα πρέπει να συμβεί, να γίνει το ένα και το άλλο και το ίδιο κάνουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, στην Επιτροπή μας τελικά να ασχολούμαστε γύρω, γύρω στο περιβάλλον του ΠΟΕ χωρίς τελικά να αγγίζουμε την ουσία των θεμάτων. Ε, τώρα, όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, πού θα δώσετε έμφαση εσείς ως Προεδρία του Συμβουλίου και τρίτον, όπως γνωρίζετε, ε, Βεβαίω δεν είστε από τη Βαβαρία, αλλά υπάρχει πολύ στενή επαφή μεταξύ Βαβαρίας και Αυστρίας. Και θέλετε μία Ευρώπη, είπατε, η οποία να παρέχει προστασία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό το σύνθημα αυτό και μια Ευρώπη η οποία μας παρέχει προστασία είναι μια Ευρώπη η οποία δεν θέλει να συμπεριλάβει στους κόλπους της, τους πάντες. Λέτε, θέλουμε εμπόριο, για περισσότερη οικονομία, άρα καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες μας. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και πολύ καιρό να ενισχυθεί το εμπόριο νότος-νότος. Οι φτωχότερες ε, περιφέρειες, οι οποίες θα πρέπει καταρχήν να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις Έχετε μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί κάτι τέτοιο, η ενίσχυση του εμπορίου νότος προς νότο. Ε, αυτή στιγμή, ε, από τότε που ασχολούμαι εγώ με την πολιτική εμπορίου, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, πλανάτε αυτό το φάντασμα, αλλά χωρίς να παίρνει πόσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Μορέλ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Τα λόγια σας ήταν ενδιαφέροντα, κάπως γενικόλογα και ίσως το καλύτερο θα ήταν να μπούμε περισσότερο στην ουσία του προβλήματος με συγκεκριμένες ε, προτάσεις γιατί βρισκόμαστε σε μια εμπορική συγκυρία αρκετά συγκεχημένη με αλλαγή στους σχετισμούς δυνάμεων και υπάρχουν πολλοί πολίτες μας που ανησυχούν. Το πρώτο θέμα που μας ανησυχεί είναι προφανώς η κατάσταση ε, των διατολικών σχέσεων. Ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε να εφαρμόζει την ε, προστατευτική του ατζέντα. Υπάρχουν ε, ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα που αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση στην εκεί αγορά, αλλά με έναν σεμνό, ταπεινό τρόπο. Το θέμα είναι κατά πόσο η Αυστρική Προεδρία τι θα κάνει όσον αφορά, για παράδειγμα, την αύξηση του κόστου των τελωνικών δασμών για τα αυτοκίνητα κάτι που για μας είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι είδους αντίμετρα μπορούμε να φανταστούμε, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει σεβαστή. Αλλά ποια είναι τα μέσα ε, μέσα στα οποία θα πετύχουμε κάτι τέτοιο. Και κάτι άλλο, όλοι ξέρουν το πολυμερές ε, σύστημα. Όλοι λένε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί ο ΠΟΕ, αλλά Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε. Ε, δεν είναι μόνο η ΕΠΑ που απονομεύουν τον ΠΟΕ. Έχει υπάρξει και άλλο πρόβλημα ε, σε σχέση με την είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ. Μια Κίνα η οποία δεν σέβεται τις συνθήκες και που τα πράγματα εδώ δεν βελτιώνονται. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, της Κίνας όπου γίνεται ξεκάθαρο το κράτος παρεμβαίνει στις εθνικές ε, αγορές Άρα οι κανόνες του ΠΟΕ δεν ε, γίνονται σεβαστές στην Κίνα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ώστε να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο είπα, όσο και η Κίνα προκειμένου να βρούμε έξυπνε λύσεις. Τρίτον, μιλήσατε για τις ε, άμεσες ε, ξένες επενδύσεις, το FDI. Ε, εδώ θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Τι σημαίνει ισορροπία. Αν θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα χαλαρό, μαλθακό κείμενο, ε, σε τι μας εξυπηρετεί. Τώρα, αναφέρατε το Βιετνάμ, τη Νέα Ζηλανδία κλπ. Ο ακτιβισμός της Επιτροπής ε, σε σχέση με τις νέες χώρες, για παράδειγμα η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, εξέρουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε εμπορικέ σχέσεις με χώρες που βρίσκονται δεκάδες, ε, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρων μακριά. Ε, ποιο είναι το όφελος. Γίνεται πιο συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε. Κυρία Σχάκη, μια από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας σωστά επισημάνατε νομίζω τα πόσα διακυβεύονται και πόσα είναι επιτάπητος και υπάρχει τώρα μια ευκαιρία επί της δικής σας προεδρίας να γίνει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για το τι σημαίνει πολυμερές εμπόριο με κανόνες γιατί και στη δική σας ε, τη χώρα βλέπαμε διαμαρτυρίες κατά των ε, τεχνοκρατικών εξηγήσεων του γιατί έχει σημασία το εμπόριο. Και τώρα είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο και νομίζω ότι θα πρέπει να αγκαλιάσετε και εσείς το θέμα του εμπορίου με κανόνες και πώς μπορεί να ε, τους ωφελήσει όλους ως ε, μια σημαντική υποτεραιότητα. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ανέφερε και ο πρόεδρος, ο έλεγχος εξαγωγής των αγαθών διπλής χρήσης. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό και νομίζω ότι καταλήξαμε τελικά σε μια στιβαρή θέση που εισάγει νέου ελέγχου για τεχνολογίες παρακολούθησης που μπορεί να επηρεάσουν πολύ την κυβερνοασφαλεία αλλά και τα δικαιώματα των ανθρώπων ε, οπουδήποτε στον κόσμο και τώρα η πτυχή των δικαιωμάτων και αυτή πρέπει να αξιολογείται πριν δοθεί μια άδεια τους εξαγωγείς και δυστυχώς ε, δεν κινήθηκε το θέμα από την Βουλγαρική Προεδρία οπότε αναμένουμε από εσάς να βρείτε μια θέση στο Συμβούλιο και να πάμε σε τριμερή διάλογο γιατί αν δεν γίνει τώρα θα είναι μια χαμένη ευκαιρία και εμείς ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε που μπορούμε για να προχωρήσει το θέμα αυτό και να καταλήξουμε σε μια όσο δυνατόν ευρύτερη συνένεση. Οπότε καλή τύχη εύχομαι και αναμένω την συνεργασία με την Προεδρία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. τότε περνάμε στην Γκουέ και τον Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας και μάλλον υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα επιτόπιτος και για νομοθεσία και για της ε, διμερής ε, σχέσεις στο Συμβούλιο, άρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε η ότι πρέπει να σκεφτούμε το πολυμερές ε, εμπόριο και ειδικά η Αυστριακή Προεδρία πρέπει να το κάνει αυτό δεδομένων και των συζητήσεων που γίνονται στο εσωτερικό της Αυστρίας για την αποφυγή των αιτίων των συγκρούσεων και μια αλληλεγγύη με τις άλλες υπήρους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο όταν μιλάμε για τον ΠΟΕ να τονίζουμε την αρχή του δίκαιου εμπορίου. Εδώ πέρα ακριβώ θα με ενδιαφέρε να μάθω τι θα κάνετε εσείς συγκεκριμένα το επόμενο εξάμεινο. Δηλαδή συνεργασία για τους κανόνες και ρυθμιστική συνεργασία. Ε, συνεργασία με τις ΙΠΑ και την Κίνα. Η Κίνα έχει κάνει κάποιες προτάσεις και ήδη στο πλαίσιο και των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ έχετε πει ότι και τα άλλα καρτιμέλη του ΠΟΕ πρέπει να συνεργαστούν στενότερα και ήδη ιδίω όσον αφορά την ευρωπαϊκή παραγωγή αυτοκινήτων παρά τους ε, τιμωρητικούς ε, δασμούς ε, στην Κίνα υπάρχει το θέμα του τι γίνεται με τις ΙΠΑ δεύτερον για τις διμερείς συμφωνίες πρέπει να διαπραγματευτούμε την συμφωνία Μερκοσούρ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και στον ΟΗΕ όσον αφορά την αδειοδότηση ζυζανιοκτώνων από την Βραζιλιανική Εθνοσυνέλευση. Θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος να υπονομευτούν κάποιες προδιαγραφές. Τρίτον, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ε, θα πρέπει να εστιάσουμε σε μια διαμόρφωση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Για το, πολιετές, ε, το πολυμελές με το δικαστήριο δεν είπατε τίποτα. Δεν ξέρω, θα κάνει κάτι σχετικά η Αυστριακή Προεδρία. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Ντάτμοθ για το EFTD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο πράγματα στις ΙΠΑ και τους δασμούς αυτοκινήτων. Λέει εδώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία πως ε, η ΕΠΑ είχε ένα εμπορικό έλλειμμα 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως εγώ δεν πιστεύω στον μερκαντιλισμό που ήταν μια γαλλική ιδέα επινόηση του Κολμπέρ, μεγάλου Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι ο πρόεδρος των ΙΠΑ πιστεύει στον μερκαντιλισμό δεν ξέρω εάν θεωρεί ότι είναι διάδοχος του Κολμπέρ, ε, τουλάχιστον όχι με αυτά τα λόγια, αλλά πιστεύει στα εμπορικά ισοζύγια. Οπότε στην συζήτηση αυτή ε, για τις ΙΠΑ, το πλαίσιο το οποίο δεν αναφέρεται είναι το ότι οι ΙΠΑ έχουν μεγάλο ε, έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για το θέμα των αυτοκινήτων που ανέφερε ο συνάδελφος, πρέπει να επισημάνουμε ως γεγονός ότι οι δασμοί των ΙΠΑ ε, για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα είναι 2,5%. Οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα είναι 10%. Οπότε αν είναι να αρχίσετε να φωνάζετε ότι οι ΙΠΑ ε, συμπεριφέρονται σχρά και προστατευτικά, κάτι με το οποίο συμφωνώ, μια καλή αρχή θα ήταν να γίνει κάτι για να μειωθούν τουλάχιστον οι ευρωπαϊκοί δασμοί στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Ε, και θα ήθελα να σας το προτείνω ως προτεραιότητα για την Προεδρία σας το έλλειμμα είναι στην πλευρά των αγαθών, όχι των υπηρεσιών. Μάλιστα. Τέλος, η κυρία Ζαμέ, όχι. Δεν έχω ερωτήσεις Υπάρχουν πολλά θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι για το γάλα, για την ε, γεωργία κλπ. Υπάρχουν, υπάρχει συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το θέμα είναι ποια μέτρα θα λάβει η Αυστρακή Προεδρία με τη ΣΥΠΑ. Είναι ένα θέμα που ανέφεραν επίσης οι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο για μένα είναι επίμαχο είναι η προσέγγιση της Αυστρίας ε, σε, στη σχέση Ανατολής-Δύσης. Ε, και αυτή η νέα προσέγγιση με το δρόμο του μεταξιού ε, νομίζω ότι δεν πάει, δεν βαίνει σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό. Για τους πράσινους, ο κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κυρία Υπουργέ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Η πρώτη σχετίζεται με αυτό το οποίο ανέφερε ο Χέλμουτ Σόλτς, το δίκαιο εμπόριο. Γνωρίζετε ότι έχει δυσκολίες στο εμπόριο που οδηγούν στην φυγή ανθρώπων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έτσι μπορούμε να λύσουμε προβλήματα της Ευρώπης. Ε, Αυτή τη στιγμή η αλλαγή της συμφωνίας με το Μαρόκο, ας πούμε, λόγω της Δυτικής ε, Σαχάρας. Αν μπορείτε να μας κάτι σχετικά. Η άλλη μου ερώτηση είναι εξής θα ασκήσετε μια πιο ενεργή πολιτική απέναντι στην Κίνα και την ε, Ρωσία που τα έχουμε λίγο κάπως ως ε, αποπέδια στο εμπόριο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και τρίτον, το είπε και ο κύριος Πρόεδρος, τι γίνεται με την ε, διπλή χρήση. Για μένα δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να χρειάστηκε τον διπλάσιο χρόνο και να μην κατέληξε τελικά σε μια γνωμοδότηση σε σύγκριση με το Κοινοβούλιο. Μόλις ε, ε, έλαβα μια επιστολή από την αντιπροσωπεία σας εδώ στις ε, Βρυξέλλες, πιθανώς την γνωρίζετε, ότι δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά. δεν μπορούμε νομίζω να το δεχτούμε έτσι απλά. Ε, είναι, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είπατε ότι το σύνθημα της προστασίας σας θα είναι η προστασία. Αυτή, δεν αφορά όμως μόνο εμάς σε αυτήν την αίθουσα, αλλά και ανθρώπους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, εάν συνεχίσουμε έτσι. Σε αυτήν την περίπτωση δεν περάσει. Ο... Στην περίπτωση του δεν θα περάσει ο θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαπραγματεύσεις. Σας παρακαλώ να το έχετε κατά αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχετε τώρα 10 λεπτά για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Για το θέμα είπα Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου χωρίς να ξεχνάμε και τα ζητήματα διπλής χρήσης τα οποία θα αναφερθώ. Το βασικό είναι ότι οπωσδήποτε ο ΠΟΕ είναι ένας οργανισμός τον οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές για τη μετασχηματίζεται η οικονομία, οι εμπορικές σχέσεις και οι φίλοι μας δεν είναι αυτοί που ήταν στο παρελθόν Γι' αυτό σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως προς αυτό. Εμείς ανησυχούμε λοιπόν πάρα πολύ, ανησυχούμε σοβαρά στο Συμβουλίο για την συμπεριφορά των ΙΠΑ και θα προσπαθήσουμε ε, με την Κομισιόν να την επηρεάσουμε, αλλά είμαστε και ρεαλιστές ε, στο πλαίσιο της ε, λήψης αποφάσεων από την άλλη πλευρά. Αν δούμε το παρελθόν, ξέρετε ότι η εισαγωγή των δασμών ε, δεν ωφέλησε ποτέ στο παρελθόν και επί Μπούς ε, του πρεσβύτερου και επί Ομπάμα επί αυτών των παρέντων ε, επιβλήθησαν δασμοί και στα ελαστικά και σε άλλα πράγματα τα οποία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις μας, ε, τότε θα πρέπει να δούμε και την εποπτεία των διαπραγματεύσεων ε, και βεβαίως για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών να ρίξουμε λίγο περισσότερο βάρος και έχουμε κάποιες ιδέες που έχουμε αναφέρει ήδη. Μία ιδέα είναι να έχουμε πιο ευέλικτες διαπραγματευτικές εντολές. Όπως είδαμε στο Buenos Aires η ομοφωνία είναι μια πρόκληση. Θα μπορούσαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να σχηματίσουμε κάποιες ομάδες ε, πυρήνα θα έλεγα που θα μπορούν μετά να διευρυνθούν και οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούμε έτσι και στον ΠΟΕ. Επίσης πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για τις επιδοτήσεις ε, της βιομηχανίας, για την πνευματική ιδιοκτησία να βρεθεί μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη και την διαφοροποίηση των αυξομενών χωρών. Δεν είναι δυνατόν η Κίνα να κρύβεται τώρα πίσω από την ταμπέλα της αναπτυσσόμενης χώρας. Πρέπει να έχουμε κάποια πιο αναπτυσ... κάποιον πιο αποτελεσματικότερο μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και υποπτία. Είναι μια διαδικασία όμως που πρέπει να κινηθεί και από τις δύο πλευρές και από τα κράτη-μέλη και εδώ πέρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ε, να παίξουμε τον κύριο ρόλο αλλά και από τον ΠΟΕ τον ίδιο πρέπει να έρθουν κάποιες ιδέες ε, και να προχωρήσουμε και να υπάρξει κάποια διασφάλιση. Για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εισαγωγή δασμών σε χάλιβα και αλουμίνιο. Νομίζω ότι αντιδράσαμε μετρημένα αλλά ξεκάθαρα. Γενικώ βεβαίως η επιβολή δασμών και από πλευράς μας μας γυρίζει πίσω και θα γυρίσει μπούμεραγκ τελικά. Εντάξει, ήταν λίγο αστείο το θέμα με τη Harley Davidson, αλλά αμέσως ανακοίνωσε η Harley Davidson ότι θα μεταφέρει θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, οπότε θα πρέπει ακριβώς να είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρξουν άλλες απειλές για δασμούς στα αυτοκίνητα να αντιδράσουμε ένα ανάλογο πακέτο. Το πρώτο πακέτο δεν περιέχει μόνο την Harley Davidson, τα Levi's κτλ. αλλά και προϊόντα χάλιβα και γεωργικά. Αν έρθει πακέτο θα πρέπει να φτιάξουμε και εμείς ένα άλλο πακέτο αλλά βεβαίως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ της Ευρώπης και των άλλων χωρών και θα πρέπει ακριβώς να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το οποίο είπε η Ένωση των Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών ότι ε, μπορεί να ανταποκριθεί με μηδενικούς δασμούς. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τους μηχανισμούς ε, του ΠΟΕ. Θα πρέπει ακριβώς ε, να χρησιμοποιηθούν μόνο από τις Ίπα, Θα πρέπει να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις για να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, για το θέμα της ανάπτυξης ε, και μιας ισορροπημένης ε, εμπορικής ε, πολιτικής οπωσδήποτε θα στηρίξουμε αυτό το κεφάλαιο της αηφορίας. Για εμένα οι κυρώσεις δεν είναι το κατάλληλο μέσο. Ο στόχος μας είναι να διαμορφωθούν κάποιες ε, εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα είναι ποιοτικέ, έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα εμπόριο το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε και προδιαγραφές, προδιαγραφές ποιοτικέ όσον αφορά τα τρόφιμα, την κτηνοτροφία σε άλλες χώρες που θα μπορούν να εξάγουν σε εμάς μόνο εάν ανταποκρίνονται σε αυτές. Τι άλλο ήθελα. Αν ναι, έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων τι εννοούσα εδώ όταν λέω ισορροπημένες. Αυτό δεν είναι κάποια απειλή. Βεβαίω οι χώρες εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές θέσεις και υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είναι ε, ξεκάθαρο εδώ ότι θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο είναι η παρακολούθηση, να δούμε τις εξελίξεις ε, και μετά να μπορέσει να γίνει μια ανταλλαγή. Κοίταξτε, εγώ είχα και 22 χρόνια εμπειρία στον τομέα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, όπου είχα δει και μεγάλες επενδύσεις και αλλού βεβαίως στον τομέα της υφαντουργίας ε, γίνονται μεγάλες επενδύσεις από την Κίνα. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανοιχτή ή να κάνει εμπόριο με όλους. Πρέπει να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό και συνδυασμό των διαφόρων θέσεων και βεβαίως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να προωθήσουμε τον έλεγχο ο οποίος δεν θα παρεμβαίνει σε ζητήματα επικουρικότητας η κάθε χώρα και η κάθε εταιρεία θα λαμβάνει τις αποφάσεις αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να γίνει ένα πρώτο βήμα για το θέμα της διπλής κρίσης ένα σημαντικό θέμα. Είδαμε και ακούστηκε η κριτική σας ε, γιατί δεν υπήρχε κάποια απάντηση από τους βουλγαρούς συναδέλφους. Βεβαίως Έχουμε ήδη 10 Ιουλίου και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει το θέμα. Έχει γίνει η προεργασία και οπωσδήποτε δούμε και την αποτελεσματικότητα και την συνοχή του συστήματος στρατηγικών εξαγωγών. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως είναι ταυτόχρονα και αυτό αφορά και τις δύο πλευρές και τον ανταγωνισμό και την, το ε, νόμιμο εμπόριο των αγαθών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ε, εξάγεται ένα πυροσβεστικό όχημα σε κάποια χώρα, πολλές χώρες ε, αποφασίζουν μεμονωμένα ανασύμβαση ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λαμβάνονται γενικές αποφάσεις αλλά μόνο κατά περίπτωση και πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία κάποιων χωρών που έχουν εργαστεί πάνω στο θέμα. Είναι ένα σχετικά περίπλοκο ζήτημα. Ακούγεται απλό αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει να εξετάζουμε πολύ προσεκτικά και αυτό θα κάνουμε και βεβαίως ε, θα είμαστε σε επαφή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτούς τους έξι μήνες. Δεν μπορώ να σας ε, πω τώρα κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά οπωσδήποτε θα παρέμβουμε όπως κάναμε και σε 9 Ιουλίου. Μερκοσούρ και εμπορική συμφωνία. Ένα σημαντικό σημείο της συμφωνίας αυτής και των συμφωνιών είναι να είναι ποιοτικές ακριβώς ε, για να φέρουμε και τις προδιαγραφές μας σε άλλες ε, χώρες, ε, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης και για τον Μερκοσούρ νομίζω υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά που δεν αφορούν μόνο το θέμα της γεωργίας αλλά και ζητήματα προϊόντων για εμάς λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα διαφάνειας Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατάσταση δίκαιη και έχει μεγαλύτερη σημασία η ποιότητα από την ταχύτητα και θα δούμε το τι θα ε, λάβουμε ως μηνύματα τις επόμενες ημέρες και γνωρίζω βεβαίως ότι πρέπει πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την συνεργασία από την άλλη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. εάν η βραδύτητα είναι ένδειξη για την ποιότητα μιας συμφωνίας, τότε η συμφωνία αυτή η Μέρκοσούρ θα είναι η καλύτερη δυνατή γιατί τη διαπραγματευόμαστε εδώ και 20 χρόνια. Τώρα υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι και θα έλεγα 20 λεπτά να βάλουμε σαν ε, πλαίσιο ha già risposto la Ministro, che auguro, a cui auguro buon lavoro. Λοιπόν, κοίταξτε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο εξάμεινο αυτό και ελπίζω να κλείσετε πολλά θέματα, όχι μόνο τον διεθνή, αλλά όλα. Λοιπόν, μια ερώτηση τώρα. Και σας ευχαριστώ για την απάντησή σας για την ε, Ρωσία. Οι κυρώσεις ε, ανανεώθηκαν στο τελευταίο συμβουλίο για άλλους έξι μήνες. Τι ε, στάση θα κρατήσετε απέναντι στην Ρωσία σε σχέση με το εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και θερμά συγχαρητήρια που επικρόσετε τη ΣΕΤΑ. Δυστυχώ η Γερμανία δεν το κατάφερε ακόμα, το κατόρθωσε, αλλά το προσπαθούμε. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία αφορά το ζήτημα της εξαπιστίας και του εμπορίου. Σε ποιο βαθμό εσείς και η κυβέρνησή σας θα δεσμευθείτε στο πλαίσιο της Προεδρίας προκειμένου να διατηρήσετε τον ευρωπαϊκή, ε, να προστατεύσετε την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ζώνη ελεύθερου εμπορίου και να εξασφαλίσετε το χώρο Schengen ως χώρο διακίνησης ε, προϊόντων, εμπορευμάτων. Το άλλο θέμα αφορά την ε, καταπολέμηση των αιτίων εξόδου από την Αφρική. Εδώ η Κίνα έχει αναλάβει ενεργό δραστηριότητα. Αυτό δεν το κάνει από ανθρωπισμό, αλλά λόγω των οικονομικών της συμφερόντων. Σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να συνοδευτεί από μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Αφρική. Ακριβώς σε διασύνδεση με την καταπολέμηση των αιτίων φυγής των πολιτών αυτών των χωρών, ούτω ώστε οι άνθρωποι εκεί να έχουν μια οικονομική προοπτική να παραμείνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο... Κύριε Περέρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε σε αυτή την Επιτροπή. Ε, καταρχήν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιον ρόλο αποδίδεται στην εμπορική πολιτική ως εργαλείο πρόσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφερθήκατε στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς σκέφτεσαι να εγγυηθείτε την εφαρμοσιμότητα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυνατόν να εκπονηθεί ένας μηχανισμός που βασίζεται σε κυρώσεις, επιβολή κυρώσεων. Δεύτερον, πώς αξιολογείται την κατάσταση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus ε, ε, σε σχέση με την κατάσταση των χωρών της Αφρικής. Τώρα, όσον αφορά την εμπορική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς αξιολογείται όσον αφορά την δεσμευτική συνθήκη και τη θέση των Ηνωμένων Εθνών να εκπονήσουν ένα σύστημα το οποίο να υποχρεώνει τους πολυεθνικούς ε, ομίλους και τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των θεμελιωδών ε, αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, θα ήθελα να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση όσον αφορά την ανανέωση της συμφωνίας με το Μαρόκο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε κατά νου, ούτως ώστε να μπορέσετε να επιλύσετε ε, τα ζητήματα των εμπορικών και λευτικών συμφωνιών με το Μαρόκο. Επίσης, προσυπογράφω όσο είπε ο κ. Δάντε, για το του σε σχέση ε, με την τοποθέτησή σας για τη σχέση με τη Ρωσία. Τώρα, επίσης, όσον αφαιρθεί αναφερθήκατε στις απαντήσεις σας σε κάποιους ε, στόχους που θα έπρεπε να ε, εκπληρωθούν σε σχέση με το ΠΟΕ. Ε, πώς όμως μπορείτε να εξασφαλίσετε την εδραίωση του ρόλου του ΠΟΕ. Ο Αλεξάνδρ Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Υπουργέ Σάμπρουκ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, ήδη όμως αρχίσατε, ε, απαντήσατε στην ερώτηση για τη σχέση μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ. ΕΕ. Θέλω όμως να υπογραμμίσω το ρόλο του Κοινοβουλίου και ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για την προσέγγιση προς τη ΣΥΠΑ και τον ΠΟΕ. Να προσθέσω στα σημαντικά ερωτήματα που ε, ήδη ετέθησαν ότι είστε υπεύθυνοι Υπουργό για τι ψηφιακέ υποθέσει και θα ήθελα να ξέρω πώ θα εργαστείτε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εμπορικέ πολιτικέ και συμφωνίε θα είναι πιο ευθυγραμμισμένε με την ψηφιακή εποχή. Για παράδειγμα, τι ε, ροέ δεδομένων ω κομμάτια των νέων εμπορικών συμφωνιών, καθώ και τα παραρτήματα εισαγωγή ε, εισαγωγικά μάλλον παραρτήματα, οποτεδήποτε είναι αυτό δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Προύστο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που είστε εδώ και χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω στον πρώτο τριμερή σε λίγο για τις επενδύσεις. Αυτό δείχνει την εμπλοκή της Αυστριακής Προεδρίας σε αυτό το θέμα και είναι αλήθεια ότι η δική σας Προεδρία είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η τελευταία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εξού και το ενδιαφέρον να προχωρήσουμε σε διάφορα θεμελιώδη ζητήματα. Είναι αλήθεια και ο συνάδελφος μίλησε για ισορροπία. Διαπιστώνουμε ωστόσο και κατανοώ ότι για σας η Ευρώπη που προστατεύει είναι βασικό βασικός άξονας ε, της πολιτικής σας. Έχουμε, πιστεύω, μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σηματοδοτήσει το τέλος της ευρωπαϊκής ε, <laughs> Αφέλεια μέσω των ε, διαφόρων μέσων άμυνα, φιλτράρισμα και επενδύσεις σε τελευταίο εξ αυτών, αλλά διαπιστώνουμε με μια πιο έντονη βούληση του Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο και θέλω να έχω την αίσθησή σας από αυτού και έπειτα για αυτή την αίσθηση των ελευθέρων συναλλαγών, που είναι μάλιστα ένα όρο που σήμερα γίνεται πολύ άσχημα αντιληπτό από τον κόσμο. Δίκαιε συναλλαγέ, θα έπρεπε να λέμε καλύτερα, γιατί πήρα από τι ελεύθερε συναλλαγέ ε, έχουν την εντύπωση ότι πρόκειται για άγριο ελευθερισμό, ε, ενώ είναι το αντίθετο. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Μαζί με το Συμβούλιο προετοιμάζεται με το μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Όμως ε, η υπογραφή των ε, συμφωνιών είναι σημαντική, αλλά ο σεβασμός αυτών των συμφωνιών είναι ακόμα καλύτερα. Μήπω προβλέπετε, προβλέπετε αρκετά συνεπής ε, μεγάλος, δηλαδή προπολογισμό στην DG13, ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και η υπογραφή τους, που θα πολλαπλασιαστούν, γιατί αναφερθήκατε σε, και σε άλλες ε, και είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετοί να υπάρχει αρκετό προσωπικό. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία να υλοποιηθεί κιόλα. Και έπειτα αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη. Γιατί αν θέλουμε η Ευρώπη να γίνεται σεβαστή, θα πρέπει το σύνολο των κρατών να είναι αλληλέγγυα όταν επιβάλλονται κυρώσει. Γιατί διαφορετικά τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν αντίκτυπο. Ευχαριστώ, κυρία Χάιντς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να με συγχωρέσετε, αλλά η καθυστέρησή μου οφείλεται στο γεγονό ότι είχα κάποιες... Ε, έπρεπε να παραστώ σε μια άλλη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Μεταφορών. Λοιπόν, η εμπορική πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ευημερίας, αλλά θα πρέπει να είναι δίκαιη και θεμητή. Εδώ συμφωνούμε όλοι. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε το εμπόριο για όλους. Αυτό για μένα σημαίνει ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, και την εργοδοσία αλλά και το περιβάλλον. Πρόσβαση στην αγορά και απελευθέρωση των αγορών και, αυτό είναι και αυτά είναι σημαντικά θέματα έχω την εξή ερώτηση. Θα δεσμευτείτε με το Συμβούλιο για την βιώσιμη ανάπτυξη σε συνάρτηση με μια επιβολή κυρώσεων. Η Γαλλία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θα κάνετε εσείς τώρα. Γιατί όλα τα κεφάλαια υπόκεινται στο μηχανισμό διαιτησίας, αλλά όχι το κεφάλαιο για την βιωσιμότητα. Ε, τώρα, όσον αφορά την, ε, τις συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη, ε, δεν έχουν επικαιρωθεί εδώ οι κανόνες του ILO ε, πρόκειται να αξιολογήσετε θετικά τις ε, συμφωνίες αυτές, αν οι δύο χώρες επικυρώσουν αυτές τις συμφωνίες. Τώρα, όσον αφορά τη ΣΕΤΑ και το δημοψήφισμα, έχει εξαγγελθεί ότι ε, ένα τέτοιο δημοψήφισμα εσείς μπορείτε να φανταστείτε κάτι τέτοιο για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να στηριχθούν σε δημοψηφίσματα και αν όχι γιατί. Ένα άλλο θέμα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην εμπορική συμφωνία, ε, την εμπορική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Ε, ε αυτό θα σημαίνει ότι ε, Επίση, συμφωνείτε με το γεγονό ότι προπαιτείται η συγκατάθεση όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο κύριο Αλαφράγκα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, επίση. Σας εύχομαι καλή τύχη για την ε, θητεία της Προεδρίας σας και θα ήθελα να θέτω έμφαση σε, στα εξή θέματα. Ότι περνάμε από μια... θα πρέπει να περάσουμε από μια προστατική Ευρώπη σε μια Ευρώπη η οποία παρέχει προστασία. Το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να σα υποβάλω ευθυγραμμίζεται με τη ε, συνάδελφο που προηγήθηκε το κομμάτι που αφορά το Συμβούλιο, γιατί υπάρχει και ένα τμήμα, το οποίο, ένα μερίδιο το οποίο αναλογεί στην Επιτροπή. Αλλά υπάρχει και ένα μερίδιο του Συμβουλίου σχετικά αφορά τις συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Μεξικό. Θα επιταχύνετε τις ε, περιόδους ούτως ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας σας να προχωρήσει σε μία επικύρωση τουλάχιστον του ενωσιακού κομματιού. Τώρα, όσον αφορά ε, τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Μερκοσούρ, εδώ και πολλά χρόνια βρισκόμαστε υπό διαπραγμάτευση και υπάρχουν δύο συμπεράσματα τα τελευταία Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Στο τελευταίο ζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει διαπραγματεύσει που βρίσκονται υπό εξέλιξη και όλοι επιθυμούμε μια φιλόδοξη και εξορροπημένη διαπραγμάτευση. Το πολιτικό τμήμα της διαπραγμάτευσης έχει ήδη ολοκληρωθεί. Γι' αυτό ελπίζουμε, κυρία Υπουργέ, να κινητοποιήσετε όλες τις δυνάμεις σας όσον αφορά ε, την ολοκλήρωση ε, της διαπραγμάτευσης με τους 28 γιατί πρόκειται για μια δυσχερή συγκυρία. Έχουμε τις ε, εκλογές αυτό το χρόνο στη Βραζιλία και έχουμε τις εκλογές τον επόμενο χρόνο στην Αργεντινή. Θα υπάρξει μια ισορροπημένη λύση σε όφελος για των πολιτών μας. Κυρία Υπουργέ, και από τη δική μου πλευρά, τρία σημεία. Ακούσαμε πολλά για όλες τις δυνατές, για όλες τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά η συμφωνία με την Κολομβία και το Περού δεν έχει επικυρωθεί από την Αυστραλία. Από την Αυστρία, συγγνώμη. Πώς θα τοποθετηθείτε εσείς εδώ. Δεύτερον, ε, οι διαπραγματεύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο σε σχέση με την Ουγγαρία και την συμμετοχή σε διεθνείς ε, συμφωνίες, πρόσβαση σε έγγραφα και ανταλλαγέ. Εμείς θέλαμε να πετύχουμε συμφωνία με την Ουγγρική Προεδρία, αλλά το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να το κατορθώσει. Τώρα υπολογίζουμε στην Αυστρική Προεδρία να πετύχει μια συμφωνία, γιατί δεν θα ήταν καλό αν στο τέλος της ε, θητείας ε, ως ε, Κοινοβούλιο να αναγκαστούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, σας εμπιστευόμαστε ότι θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο θέμα αυτό χωρίς να απαιτηθεί αυτή η προσφυγή. Τρίτον, ποιο είναι το δικό σας μέτρο για μια πετυχημένη αυτική προεδρία Πού βάζετε το γνώμονα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην στοχοθεσία μας. Μία Ευρώπη η οποία παρέχει προστασία έχει τρεις ε, πτυχές. Το κλασικό κομμάτι της προστασίας, το οποίο συνθέτει με τους άλλους συναδέλφους, ένα κομμάτι ψηφιοποίησης, που είναι ξεκάθαρο ψηφιοποίηση για την προστασία της ευημερία και των θέσεων απασχόλησης και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για μας και το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ, το θέμα της σχέσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στο πλαίσιο αυτό είχαμε μια συνδιάσκεψη στη Βιέννη όπου ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της ψηφιοποίησης και το θέσαμε στο επίκεντρο. Και εδώ ο στόχος μας και είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τα Δυτικά Βαλκάνια, περισσότερο εμπόριο, αύξηση της εσωτερικής αγοράς, περισσότερες δυνατότητες επένδυσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αυτή την ε, συγκεκριμένη εσωτερική αγορά. Τώρα, για τις ερωτήσεις σας όσον αφορά τη Ρωσία, θα ξεκινήσω με αυτήν. Από τη δική μας πλευρά, η επιβολή κυρώσεων δεν είναι αυτό σκοπός. Και ως Αυστρία πάντοτε πραγματευθήκαμε το θέμα, ε, ενισχύοντας το διάλογο, υποστηρίζουμε μια ευρωπαϊκή συνένεση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, ε, ε, και στη συνέχεια μια σταδιακή προσαρμογή. Αλλά βεβαίως ε, καταρχήν χρειάζεται και μια κίνηση από την άλλη πλευρά. Στο θέμα Αφρική. Εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η καταπολέμηση των αιτίων εξόδου των πολιτών από αυτές τις χώρες. Το εμπόριο είναι εδώ ένα σημαντικό εργαλείο για τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να φορτώνονται υπερβολικά με τέτοιους όρους. Ε, όσο αφορά το Μερκοσούρ είχαμε κάτι παραπλήσιο με τον Καναδά και μιλάω βάσει της μου εμπειρίας, γιατί αντιμετωπίσαμε πολύ σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο της εφαρμογής. Τώρα, με τι αλλαγέ τη ΣΥΠΑ έχει αλλάξει κάπως και η ατμόσφαιρα, το κλίμα. Το είπατε και ε, ο ίδιος. Ε, χρειαζόμαστε νέες ε, εξειδικευμένες εταιρικέ συμφωνίες που να μην είναι όμως υπερβολικά φορτωμένες. Και οι κυρώσει δεν αποτελούν ποτέ κομμάτι της λύσης κατά την άποψή μου. Θα Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε ψηφιοποίηση και εμπορικέ ροές. Σημαντικό εδώ είναι να δώσουμε έμφαση με το κομπέτ στην ψηφιοποίηση, βιομηχανοποίηση, ανά βιομηχανοποίηση της Ευρώπης, τεχνητή νομοσύνη, ρομποτική κλπ για να ξαναφέρουμε πίσω επιχειρήσεις που έχουν μετεκατασταθεί και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση. Όλα αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μου, στο πλαίσιο του ΚΟΜΠΕΤ. Έχετε θέσει και ένα ερώτημα σε σχέση με το θέμα εμπόριο και δικαιώματα των εργαζομένων και περιβάλλον. Όπως σας είπα, αυτή, το υπερβολικό φόρτωμα με όρου των εμπορικών συμφωνιών οδήγησε σε αδιαφάνεια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε διαφανεί διαπραγματεύσει. και να μην τις φορτώνουμε υπερβολικά με όρου. Τώρα, είμαστε υπέρ Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και των αντίστοιχων συμφωνιών. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται και ζητήματα προστασία των επενδύσεων εδώ μπορούμε να συζητήσουμε με, τις εμπορικές, με τους εμπορικούς εταίρους και να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας. Law making, ε, διεθνείς συμφωνίες. Στόχος μας εδώ είναι ο στι Στις 30 Μαΐου είχαμε μια πολιτική συνεδρίαση. Η Προεδρία διαβουλεύθηκε με την αντιπροσωπεία για, τα προσεχή βήματα. Χαιρόμαστε που μπορούμε να κάνουμε θεσμικές συζητήσεις. Θέλουμε εδώ να υπάρξει ένα ισορροπημένο πακέτο. Θα το υποστηρίξουμε. Κατανοούμε την επιθυμία για διαφάνεια. Αλλά και βεβαίως δεν είμαστε εδώ μόνοι αλλά υπάρχουν άλλες πολύ επικριτικές ε, τοποθετήσεις και θα πρέπει να τις ακούσουμε. Το τελευταίο θέμα ήταν ε, η υποανάπτυξη χώρες. Ήδη αναφέρθηκα στο θέμα αυτό. Το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων είναι εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τις αναπτυσσόμενες χώρες που θα πρέπει να εξασφαλίσουν μία πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό μας χαροποιεί, αλλά θα εξετάσουμε την κατάσταση και θα παρέχουμε τη δική μας υποστήριξη. Uh, um, Τώρα, όσον αφορά την Κολομβία, έχουμε επίγνωση της σπουδαιότητας αυτού του ζητήματος. Θα το εξετάσουμε. Τώρα, όσον αφορά την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, βεβαίως ε, ο καθένας μπορεί να την κάνει, αλλά δεν είναι ε, σόφελός ε, μας ή προς το δικό μας συμφέρον. Θα δούμε και εδώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν απαντήσατε όσον αφορά την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Α, και την άποψή σας για τα δημοψηφίσματα ως εργαλείο. Βεβαίως τα δημοψηφίσματα μπορούν να διεξάγονται, ο καθένας μπορεί να τα κάνει. Μπορώ να σας δω πως αξιολογώ στην συμφωνία με τον Καναδά. Είναι μια υψηλής ποιότητας, ισορροπημένη συμφωνία, ίσως και πιο αξιόλογη συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση τόσο εμείς, όσο και διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι επιμέρους χώρες, ότι δεν υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά την επικύρωση, όσον αφορά το δικαστήριο επενδύσεων το οποίο μέλει να συσταθεί. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία που έχουμε εδώ και σε συνάρτηση με τον ΠΟΕ να συσταθεί ένα δικαστήριο μόνιμο δικαστήριο για πέντε χρόνια, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τρίτες χώρες, Καναδά και λοιπά. Και αυτές θα συμμετάχουν σε σύσταση του δικαστηρίου. Έτσι όπως γίνεται και με τα εργατικά δικαστήρια, τα οποία είναι ενδεδειγμένα εγώ ως πρώην δικαστής είμαι υπέρ αυτών των λύσεων γιατί μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά βεβαίως ε, μετά από κάποιες βελτιώσεις. Όσον αφορά τις νομικές αποφάσεις, δεν ακούγεται. Α, και εδώ θα πρέπει να τις εμπιστευτούμε και αν υπάρχει μια άλλη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η απόφαση είναι εφαρμοστέα σε όλες τις χώρες. Εμείς στην Αυστρία είμαστε η 12η χώρα που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης εδώ. Κυρία Χίρς, είχα ρωτήσει σε ποιο βαθμό θα προστατεύσετε το χώρο Schengen, την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Ναι, ευχαριστώ, λέει Υπουργό, που μου υπενθυμίσετε αυτή την ερώτηση. Για μα, ε, βεβαίω, η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων είναι σημαντικό θέμα. για βασική αρχή εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Ο στόχο μα είναι ξεκάθαρο. Μια Ευρώπη η οποία παρέχει προστασία θα πρέπει να εξασφαλίσει και τα εξωτερικά τη σύνορα, ούτε ώστε στο εσωτερικό τη να εξασφαλίζονται αυτέ οι ελευθερίε. Ε, εμένα με ενδιαφέρει αυτό προσωπικά. Εγώ είμαι από το Kitzbühel, πάω από την ε, Βιέννη στο Kitzbühel και κάνω μια ώρα αυτοκινητόδρομο. Ε, θε, νομίζω πρέπει να βρούμε μια γενική λύση και εμείς ως Προεδρία θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το εξωτερικό σύνορο. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο στόχος μας ούτως ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ελευθερίες που προβλέπονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο κοινό μας έργο. Και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για να εφαρμόσουμε τα όσα συζητήσαμε σήμερα. Okay, now we... Ωραία. Περνάμε σημείο 13. Η ρήτρα διασφάλισης. Κάτι το καινούριο. Κανονικά για κάθε συμφωνία να έχουμε κάτι το σχετικό και τώρα Κομισιόν προτείνει κάτι το οποίο θα είναι οριζόντιο Εισηγητής είναι ο κύριος Φιέλνερ ο οποίος όμως ε, απουσιάζει λόγω κολλήματος και τον αντικαθιστά ο κύριος Σαλαφράνκα. Μάλιστα, όντω. Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφο δεν μπορούσε να είναι παρόν και μου ζήτησε, σαν όνομά του, να σα αναφέρω κάποια σχόλια και αντιδράσει στην πρόταση τη Κομισιόν. Ο κύριο Φέλνερ θεωρεί πω οι ρήτρε ασφαλεία για τι διμερείς ε, συμφωνίε στην πράξη είναι ένα εργαλείο απελευθέρωση και που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν ε, μία διέξοδο για περίπλοκε περιστάσει. Ε, ε, μάλιστα με βάση την πρόταση της Κομισιόν για αυτά τα μέτρα για τις ρήτρες ασφαλείας ε, ε, να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Επιστεύει λοιπόν γι' αυτό ότι πολλοί από αυτούς τους κανόνες περιλαμβάνονται ήδη στις διμερείς συμφωνίες του ΠΟΕ και επίσης στις πολυμερείς συμφωνίες. Πιστεύει και νομίζω πως έχει δίκιο πως ε, είναι ένα περιθώριο ελιγμού ε, σχετικά περιορισμένο για τον νομοθέτη. Ε, ο όμως θεωρεί ότι όταν αυτό είναι δυνατόν είναι φταίο αυτοί οι γενικοί κανόνες να ισχύουν μουτάτες μουτάντης και στις διμερείς συμφωνίες. Ο κύριος Φέλνερ λέει ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι κατά κάποιο τρόπο η μετάγραφη των διμερών συμφωνιών που υπάρχουν ήδη σε κάποιες συμφωνίες όπως αυτή με την Κορέα, τη Μολδαβία, την Κολομβία ε, και θα ήθελα ωστόσο να εκφράσει κάποιους προβληματισμούς. Λέει ότι είναι υπέρ αυτής της νέας οριζόντιας νομοθεσίας που μπορεί να καλύψει τις ισχύουσες συμφωνίες. Ωστόσο, επίσης πιστεύει πως αυτή του είδους οι ρυθμίσεις δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απαγορεύουν τη δυνατότητα ύπαρξης ρητρών ασφαλείας που υπάρχουν ήδη στις διμερείς συμφωνίες. Λέει πως αυτό ισχύει για τις συμφωνίες ε, με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Λέει επίσης ότι αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να καλύψει και κάποιους νέους μηχανισμούς, όπως ο νέος μηχανισμός ε, σταθεροποίησης για τις μπανάνες, καθώς και ο μηχανισμός ε, duty plus για την Κορέα. Ελπίζει ο κύριος Φιέλνερ ότι θα βρεθεί σύντομα συμφωνία και με τη Μερκοσούρ και αν είναι δυνατόν να υπάρχει και εκεί ένα μηχανισμό σταθεροποίηση για τα ευαίσθητα προϊόντα. Επίση αναφέρει ότι οι προβλέψει που θα συνοδεύουν αυτού του οριζόντιου μηχανισμούς δεν είναι αρκετά λεπτομερεί στην πρόταση τη Κομισιόν και επιφυλάσσεται επί τη βάση τη εμπειρία του εξυγχρονισμού των μέσων ε, ε, πορική συνεργασία, να υποβάλει κάποιε τροπολογίε στην πρόταση της Κομισιόν. Αυτά είναι τα σχόλια λοιπόν που σας υπέβαλα στο όνομα του εισηγητή του κυρίου Φιέλνερ. Ε, ήθελα να τα μοιραστεί με τους συναδέλφους και φαντάζομαι ότι στις επόμενες ε, συζητήσεις του θέματος θα μπορέσει αναλυτικά να μοιραστεί μαζί μας τις ιδέες του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thanks a lot for the Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Μαυρίδης για τους Σοσιαλδημοκράτες. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για την ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το ξαναδούμε το θέμα βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, αν ήταν εδώ ο εισηγητής, θα ήθελε να μου εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ένας μηχανισμός σταθερότητας για ευαίσθητα προϊόντα. Αλλά τούτου λεχθέντος επαναλαμβάνω πως τα μέτρα αυτά είναι αναπόσπαστο τμήμα των συμφωνιών ελευθερίου για να δημιουργηθεί σοβαρή βλάβη ή απειλή στην εγχώρια βιομηχανία ενός παρόμοιου ή άμεσα ανταγωνιστικού προϊόντος. Σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να απλοποιηθεί η διαδικασία για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης με μια οριζόντια τέτοια ρήτρα και μηχανισμό. Θεωρούμε ότι μπορεί έτσι να υπάρχει σαφήνεια και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών με το να υπάρχουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές και διαδικαστικές υποχρεώσεις. Όμως σκοπεύουμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχυθεί το κείμενο σε κάποια ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά για την ομάδα μας. Είναι ουσιαστικό να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την εγχώρια βιομηχανία και ειδικά τι μικρέ και μεσαίε επιχείρησει, αλλά και να ε, διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγέ θα συμμορφώνονται με τι ε, προδιαγραφές τη Ένωση, Παραδείγματο κάνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πρόταση τη Κομισιόν και είναι σημαντικό για εμά. είναι η εισαγωγή κάποιων προδιαγραφών εργασιακών και περιβαλλοντικών. Επίσης, κάτι το οποίο λείπει είναι το δικαίωμα της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητάει από την Κομισιόν να αναφέρει για συγκεκριμένες ανησυχίες για τις δεσμεύσεις για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Παραδείγματο χάνει αυτό αναφέρεται και στις συμφωνίες με Κολομβία, Ισημερινό και Περού. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα πρόταση δεν υπονομεύει το δικαίωμα εξέτασής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οπότε πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία μια γνώμοδότηση για να ξαναδεί την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο άρθρο 6 παράγραφο 10 αναφέρεται ότι όταν οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπλανητικές πληροφορίες η Κομισιόν θα αγνοήσει αυτές τις πληροφορίες θεωρούμε το κείμενο πρέπει να ενισχυθεί και υπό κάποιες συνθήκες θα πρέπει να ζητήσουμε κυρώσεις για τις ε, βιομηχανίες εκείνης ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που δίνει λανθασμένες πληροφορίες στην Κομισιόν. Δεν θα μπω τώρα σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες καθώς πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αναμένουμε την έκθεση του εισηγητή. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό στην επόμενη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έμα Μακλάρκιν. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας καλωσορίζει αυτή την πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το τεχνικό για να δοθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως γίνεται και στις διμερείς συμφωνίες ε, ενώ ελπίζουμε θα υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας. δικαίωση κομισιών, Κομισιόν ενέκρινε κάποια από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για διαφάνεια ετήσιες εκθέσεις και θεωρώ ότι έχουμε μια καλή βάση για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Δεν νομίζω ότι έχουμε σοβαρές ε, διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ομάδων, αλλά για τη δική μου την ομάδα είναι σημαντικό να ολοκληρώνται οι έρευνες εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν και τα μέτρα να είναι αναλογικά και να ισχύουν για περιορισμένη περίοδο και να είναι σωστά αιτιολογημένα. Καλώς και το ηλεκτρονικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. Πού είμαι. Τι έλεγα. Συγγνώμη, κάντε ένα διάλειμμα. Α, ναι, γενικά, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην επιτρέψουμε οι ρήτρε αυτές να αποτελέσουν μια μάσκα για προστατευτισμό. Πρέπει πάντα να είναι δικαιολογημένες και με ευελιξία, αλλιώς θα υπονομεύσουν τις ε, σχετικές ε, συμφωνίες. Αλλά καλωσορίζω και στηρίζω τον εισηγητή και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ Χίρση, για την Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσωρινή άρση των εμπορικών προτιμήσεων που βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις γιατί πρέπει να αποφεύγεται όπως είπε και η αίμα ο προστατευτισμός. Ναι. Πρέπει λοιπόν ε, να οδηγούμε με τραβηγμένο το χειρόφρενο, γιατί έτσι αυξάνεται η περιπλοκότητα, όπως και ο αριθμός των εμπορικών σχέσεων. Έχουμε σημαντικό αριθμό τέτοιων συμφωνιών, οπότε θα πρέπει να έχουμε απλές διατάξεις. Σημαντικό για εμάς ως φιλελεύθερους είναι το ότι εμπλέκεται και το Κοινοβούλιο, οπότε υπάρχει ε, διαφάνεια. Οπότε χαιρόμαστε για τις ε, περαιτέρω συζητήσεις και την ε, συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, David Μάρτιν. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω την πρόταση αυτή. Νομίζω λογικό είναι να έχουμε μια οριζόντια συμφωνία αντί να γίνεται αναχώρα και κατά περίπτωση, αλλά σημειώνω ότι, με πάση συμφωνεί με τα όσα έχουμε κάνει με την Κορέα και το Περού. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι η κλίμακα, γιατί ελπίζω η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και ίσως και το Βιετνάμ να ολοκληρωθούν πριν από την λήξη της ε, θητείας μας και ο χρόνος πραγματικά πιέζει και βεβαίω ε, ο Κρίστοφερ θέλει να προχωρήσει γρήγορα και τον στηρίζω. Το ερώτημα όμως που θέλω να θέσω στην Κομισιόν, εάν, εάν που ελπίζω να μην γίνει, να ε, το ολοκληρώσουμε πριν από την κύρωση, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οποιαδήποτε δεδομένα, καταγγελίες που θα γίνουν μεταξύ της κύρωσης ε, και της εφαρμογής του κανονισμό αυτού διασφάλισης θα ληφθούν υπόψη, θα μπορούμε δηλαδή να γυρίσουμε πίσω να λάβουν υπόψη τα δεδομένα. Γιατί βεβαίω χρειάζονται και έξι μήνες για να γίνει μια έρευνα, οπότε δεν νομίζω να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα το να ληφθεί υπόψη κάτι τέτοιο. Βεβαίω είναι ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, το οποίο θα απαντήσει ο κύριος Μίχελς ε, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Μάλιστα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ και γιατί προβλέπετε αυτού του είδους τη συζήτηση. Άκουγα την προηγούμενη συζήτηση όπου συζητήσατε για τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ε, για την Ευρώπη που προστατεύει και όντως ε, αυτό είναι ο στόχος των διμερών συμφωνιών ότι δηλαδή να δώσουμε προτιμήσεις στους εμπορικούς μας εταίρους αλλά εάν οι οικονομικοί μας φορείς έχουν προβλήματα πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να άρουμε αυτές τις προτιμήσεις ή να τις αναστείλουμε. Και ακριβώς αυτό κάνει αυτός ο προτινόμενος κανονισμός. Αρχίσαμε με διαπραγματευτική εντολή, δεν... Ε, προβλέπει αυτή η διαπραγμάτευση, τι θα, αυτός ο κανονισμός μάλλον, τι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στο μέλλον, αλλά Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που διαπραγματευτήκαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν μέσω και με την βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι περισσότερο διαδικαστικές πτυχές, πώς γίνονται δηλαδή οι έρευνες, πώς ε, δίνουμε τα δικαιώματα στους εταίρους να παρέμβουν και να περλάβουν εκεί και την έρευνα των συνθηκών. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, όπως είπατε πρόεδρε. Ίσως είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για έναν οριζόντιο κανονισμό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για ένα τέτοιο είδος κανονισμού. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, το έχουμε κάνει για την Κορέα, την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία, το Περού, το, το Ισημερινό, τη Γεωργία, τη Μολδαβία. Και έχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία και έχουμε επίσης ωφεληθεί από προτάσεις που έβαλε το Κοινοβούλιο στο παρελθόν, γιατί τις έχουμε δεχτεί μέσω του συγκεκριμένου ε, κανονισμού. <clears throat> Και πιστεύω πως τώρα καλό είναι να έχουμε ένα κανονισμό που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και δεν θα χρειάζεται πάντα να επαναλαμβάνουμε την ίδια προσπάθεια. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτή την εμπειρία και έπειτα αυτό που προτείνουμε είναι να ε, ανανεωθεί στο μέλλον ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέες συνθήκες. Αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν για παράδειγμα με το Μερκοσούρι χρειαστεί να έχουμε έναν μηχανισμό σταθεροποίησης για την μπανάνα. Μπορεί επίσης να γίνει αν υπάρχει κάποιο άλλο είδος μηχανισμός τον οποίο διαπραγματευόμαστε στις συμφωνίες. Η νομοθεσία δεν μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό, αντίθετα μας επιτρέπει να ε, το εντάξουμε μέσα στον κανονισμό. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι σημαντικό, αλλά το βλέπουμε περισσότερο ως μια ευθυγράμμιση της διαδικασίας επί τη βάση της εμπειρίας που έχουμε σωρεύσει. Για το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν ο κανονισμός αυτός να είναι έτοιμος όταν θα αρχίσουν ε, να ισχύουν οι συμφωνίες με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη αλλά δεν είναι και απαραίτητο γιατί για να ξεκινήσει μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να δει κανείς ποιες είναι οι συνέπειες της ε, έναρξης ισχύω της συμφωνίας και αυτό παίρνει κάποιους μήνες. Μόνο μετά από κάποιους μήνες λειτουργία ε, λειτουργίας μιας συμφωνίας μπορούμε να δούμε αν τηρείται ε, και πώς εφαρμόζεται και κατά πόσο αυτό φέρνει κόστος, επιβαρύνει με κόστος. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν ιδανικά θα πρέπει να είναι έτοιμος όταν θα αρχίσει να ισχύει και η συμφωνία, αλλά Και αν δεν το ε, καταφέρουμε, δεν θα μας εμποδίσει αυτό από το να προβούμε στις απαραίτητες ε, δράσεις. Όλα αυτά φυσικά θα τα εξετάσουμε και ελπίζω ότι όλοι μαζί, αν χρειάζεται να βελτιώσουμε τον κανονισμό, θα το κάνουμε και έτσι θα έχουμε μία σταθερή και διαφανή νομική βάση που θα είναι εύκριστη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής ο ίδιος θα κλείσει. Εγώ να συνοψίσω τη συζήτηση. Μπράβο σε όλους, καταπληκτικές οι παρατηρήσεις σας. Όχι, να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη που, ε, που άργησα. Είχα μια εμπειρία της Brussels Airlines όταν φτάνει στις 6 ας πούμε το πρωί το στο αεροδρόμιο και ακούς ένα μήνυμα που λέει ότι θα φύγει στις 9.30. Εν πάση περιπτώσει, Περιθώριο ελιγμού δεν έχουμε και πολύ, γιατί δεσμευόμαστε από την νομοθεσία ΠΟΕ, το πλαίσιο που ισχύει εκεί δηλαδή. Νομίζω πως δεν είναι και τόσο μεγάλο όμως αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά στην ουσία. Ούτε χρειάζεται να φτιάξουμε μια νέα δομή ε, ε, ασφαλιών. Απλά πρέπει να γίνει ε, οριζοντιοποίηση του συστήματος some colleagues. Οι δε καταπληκτικοί μου υπάλληλοι είπαν ότι όταν θα γίνει αυτή η οριζοντιοποίηση, αν υπάρχει τέτοια λέξη, λέει ο Μίλτης, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι να μην μετατραπεί σε προστατευτικό εργαλείο. είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το προσθέσουμε στην πρόταση της Επιτροπής. Κάποια από τα στοιχεία που είχαμε επιτυχία. όπου δηλαδή τα μέσα έχουν γίνει πιο επιτυχή και πιο διαφανή. Χάρη σε κάποιες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει να περιληφθούν, να βασιστούμε στην καλή συνεργασία και στα καλά αποτελέσματα που είχαμε. Και επ' να πω ότι προσβλέπω συνεργασία με τους συναδέλφους. Ε, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ε, κλείσαμε και με αυτό το θέμα. Διακόπτουμε και θα ε, ξαναρχίσουμε στις 2.30 εδώ στην αίθουσα την ίδια.